Καλημέρα συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε σας παρακαλώ. Can I start Ανακοινώσει του Προέδρου, αν μου επιτρέπετε να αρχίσω από αυτές. get... Πριν συνεχίσω, να σας πω τι αποφάσισαν οι συγγητές. Θα ήθελα απλώς να ενημερώσω την Επιτροπή ότι μετά από τέσσερα χρόνια εργασίας εδώ στη γραμματεία μαζί μας, μας φεύγει ο Γιάννης και πάει προς νέες προκλήσεις στη μονάδα συναπόφασης. Τελευταία μέρα σήμερα. Από τότε που ήρθε εδώ ο Γιάννης έχει εργαστεί σε πάρα πολλά θέματα, σε ένα ευρύ φάσμα ε, θεμάτων. Ξέρω ότι έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ από τότε που ανέλαβα. Θέλω να του ευχηθούμε όλοι ό,τι καλύτερο στις νέες περιπέτειες που μπαίνει στη συναπόφαση. Σίγουρα θα τον δούμε σε αυτό τον ρόλο. Γιατί από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο ποτέ δεν συμφωνεί με τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Οπότε θα τον βλέπουμε και σε αυτή τη νέα του θέση. Θα ήθελα εκ μέρους σας να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Okay. Λοιπόν, τι αποφάσισαν οι συντονιστές. Um, λοιπόν, δύο εκθέσεις. Ε, ε κανονισμός ε, για τις στατιστικές επιστροφές ε, ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές. Δεν θα εκπλαγείτε να μάθετε ότι ο πρόεδρος θα κάνει αυτή την έκθεση. Άλλη μια έκθεση για στατιστικές που του δώσατε ε, ε, πρόσφατους μήνες για τον κανονισμό για τη θέσπιση ενός προγράμματος για ε, τη ναυτιλιακή πολιτική το ΕΛΚ για τις γνωμοδοτήσεις απαλλαγή για το 2009 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης το ΕΛΚ επίσης για τη γνωμοδότηση αυτή απαλλαγέ για τους διάφορου οργανισμού ΕΜΣΑ, ΙΑΣΑ, ε, ΣΕΖΑ και Σιδηρόδρομοι Τι έχουν ενώσει όλες μαζί αυτέ σε μία γνωμοδότηση οι συντονιστέ και το αναλαμβάνουν φιλελεύθεροι. Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα δίκυκλα, τα τρίκυκλα και τα λοιπά και τα κότς η συντηρητική το ανέλαβαν η ομάδα ECR για τη γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνήσαμε να μην γνωμοδοτήσουμε για την απόφαση για λεπτομερείς κανόνες ε, για ε, το GNS. Δεν κάνουμε γνωμοδότηση αυτό. Και η Επιτροπή Ελευθεριών θα ε, κάνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη συνολική ε, προσέγγιση του ΠΙΕΝΑ για τις τρίτες χώρες, τα δεδομένα των ε, επιβατών, σοσιαλιστές και δημοκράτες θα κάνουν τη γνωμοδότηση αυτή. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα εάν η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα κάνει έκθεση για να γνωμοδοτήσουμε. Σε περίπτωση που γίνει αυτό γνωμοδοτούν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Αυτά ονόματα εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ επίσης θα ε, ε, συζητήσουμε με την Επιτροπή αυτή και θέλουμε να καλέσουμε την κυρία Χάουκ και τον εισηγητή κύριο Καρίγα Πολέντο στη συνεδρίασή μας του Νοεμβρίου για να συντάξουμε γνωμοδότηση, σχέδιο καλύτερα γνωμοδότησης μέχρι τον Ιανουάριο ε, για την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ που ξέρετε ότι είναι εξασφάλιση των οικονομικών μετά το 2013. Επιτροπολογία. Οι μόνιμοι διαρκείς εισηγητές ενημέρωσαν τους εισηγητές για μελλοντική ε, ρύθμιση ε, του προσωπικού που εργάζεται στις αεροπορικές εταιρείες. Το Δεκέμβριο μάλλον θα ε, συζητηθεί αυτό για τις εξετάσεις για τα διπλώματα ε, κυβερνητών και ερασιτεχνών. Ε, ο κύριος Αλχαντραώ είπε να το δούμε όταν έρθει στις 9 Νοεμβρίου ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΙΑΣΑ για να το συζητήσουμε μαζί. Επίσης, ενημέρωσα τους συντονιστές για το αίτημα του κυρίου Κόχλιτσεκ να τεθεί το ζήτημα των ανεμοπτέρων, γιατί τον Ιούνιο έγινε ένα δυστύχημα στην Αυστρία, θα θυμάστε. Το μέλλον των διευρωπαϊκών δικτύων των μεταφορών. Συζητήσαμε τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις και τις επιλογές και συμφωνήσαμε να επανέλθουμε στις 30 Νοεμβρίου ε, αφού θα έχουμε διαβουλευτεί στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Στα διάφορα των συντονιστών Ευρωβινιέτα ο εισηγητής έκανε μια σύντομη ανάλυση της πολιτικής συμφωνίας που ε, επετεύθη και πρότεινε να διερευνήσουμε τις δυνατότητε για περαιτέρω ε, πρόοδο κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας μετά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συμφώνησαν οι συντονιστές να γίνει αυτή η διερευνητική λοιπόν ε, κίνηση και εντολή με την προϋπόθεση να έρθει με κάποια πρόοδο να μας αναφέρει ο εισηγητής. Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με βάση το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011, οι συντονιστές αποφάσισαν να συζητήσουν στις συνεδρίες του Νοεμβρίου θέματα για πιθανή συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια το 2011. Οι συντονιστές θα έχουν έκτακτη συνεδρίαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου για να ενημερωθούμε για τη μαύρη λίστα των αερομεταφορέων, για το, την αγορά των πολιτών και τη φτώχεια μετά την δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Αυτό έχει αναβληθεί 27-28 Ιανουαρίου 2011 το έγγραφο θέσεων ε, για τις μεταφορές εγκρίθηκε στις 12 ε, του μηνός ε, με τη γραπτή διαδικασία, αλλά ζήτησε διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών να επανέλθουμε τον Ιανουάριο. Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να ενημερώσετε τους συντονιστές ποιος θα πάει στην επίσκεψη στο αεροδρόμιο του Σχίπολ στο Άμστερνταμ στις 10 Νοεμβρίου. Αν ενδιαφέρεστε, είναι ανοιχτή η επίσκεψη αυτή για όλα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών να πάρουμε να δούμε τους σαρωτές σώματος και την ασφάλεια του αεροδρομίου. Επίσης, συμφώνησαν οι συντονιστές να στείλει στον Επίτροπο επιστολή ο Πρόεδρος για τη συνέχεια που δίνεται στα ψηφίσματα ε, των, ε, του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου αποφασίσαμε κάτι στο Κοινοβούλιο, ένα ψήφισμα ε, για την πτώχευση αεροπορικών εταιριών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για μια μελέτη ε, αντικτύπου εμπεριστατωμένη και τα λοιπά, την οποία θα μας παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά πόντι. Αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για άλλα θέματα, η κυρία Λίχτεμπεργκερ και η Πράσινη έσαν το ζήτημα <laughs> της μεταφοράς μας και ε, της κυκλοφορίας στο Στρασβούργο. Αλλά είπαμε το ξανασυζητήσουμε όταν επιτέλους ψηφιστεί το χρονοδιάγραμμα για το 2012 των συνόδων στο Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επίσης μας ενημέρωσε ότι θέλουν ε, να δοθεί κάποια συνέχεια και παρακολούθηση της υπόθεσης της κρίσης με την τέφρα του ηφαιστείου και να δούμε πώς ε, θα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον τέτοια φαινόμενα σε περίπτωση που επαναληφθούν στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Έχετε ερωτήσει για όλα αυτά που σας είπα για τους συντονιστές. Εάν όχι, έχετε. Μπράιαν, πότε θα γυρίσουμε από το Σχήπολ, γιατί εκείνη τη μέρα έχουμε και μείνει σύνοδο, ξέρεις, 10 Νοεμβρίου. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε γυρίσει γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ουσιαστικά, έτσι δεν είναι. Πρέπει να γυρίσουμε στην Ολομέλεια. Στις 3 η ώρα που αρχίζει η Ολομέλεια θα είμαστε πίσω. Εντάξει. Συμφωνούμε λοιπόν και προχωρούμε. Επόμενο θέμα. Υπογραφή και σύναψη συμφωνίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καναδά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας έγκριση σχεδίου έκθεσης. ψηφοφορία είναι η έγκριση του σχεδίου απλώ. Τεστ για να δούμε δουλεύουν τα μηχανήματα. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά τώρα κάτι. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. As everybody, there's always one in the class, Michael. Has everybody voted? Ψήφισατε όλοι, πέρας. I, that's, that's okay. You can see me after class. Ωραία, μπορείς να με δεις μετά το τέλος των μαθημάτων. Ωραία λοιπόν. Πολύ καλά τα καταφέραμε. Είναι κάπως πολύπλοκος ο κατάλογος. Να περάσουμε στην ψηφοφορία, δεν υπάρχουν τροπολογίες, έχουμε μόνο την τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Τίκα. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. 29 υπέρ, κανένας κατά, καμία αποχή Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Τη απουσία της θα θέλαμε να συγχαρούμε την κυρία Τικάου. Thank you, thank you. Σε νέα ήταν η ψήφη 30 με τον κύριο Κράμερ. time the next one, So we got a 10 minute break. Διάλειμμα 10 λεπτά. Μέχρι τις 9 και μισή. Πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με συντονιστές, κυρία Πάης και ο Βαλέντε Ντελουιβέρα. Παρακαλώ, επιστρέψτε πριν από τις 9.30. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας καθίσουμε σας παρακαλώ. Θα ήθελα να, να σας εξηγήσω πώς θα προσπαθήσω να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Θα ζητήσω και από τους δύο συντονιστές να πάρουν πρώτα το λόγο για 10 λεπτά και αγαπητά μέλη. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το χρόνο αγόρευσης των συντονιστών, όπως εξάλλου είμαι και με το δικό σας χρόνο αγόρευσης. Θα περάσουμε σε ένα γύρο ερωτήσεων, θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές και τα υπόλοιπα μέλη. Όλα τα μέλη. Οι δύο συντονιστές λοιπόν και μετά το μπαλάκι σε εσάς για να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Θα επαναλάβουμε αυτή τη ε, διαδικασία μέχρι το τέλος πρωινής συνεδρίασης και το τέλος της απογευματινής. Δίχως άλλη χρονοτριβή, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω πρώτα δίνοντας το λόγο στην κυρία. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Κάρλα Πέις να πάρει το λόγο για 10 λεπτά και μετά θα μου επιτρέψει να περάσω τον κύριο Βαλέντη. recent So, it's that microphone, Carla. So, Ωραία. Κάρλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν. Αξιότιμα μέλη, θα είχα πάρα πολλά να πω για τις μεταφορές σε αυτή την πόλη. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εξηγώντας σας για ποιο λόγο ακριβώς βρίσκομαι εδώ Έχω δύο βασικά σχέδια. Το ένα αφορά τον ε, Δούναβη, τη μακροστατηγική του Δούναβη. Το άλλο θα το συζητήσουμε αργότερα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υιοθετεί μια ολιστική, μια σφαιρική άποψη. Η φετινή χρονιά συμπίπτει με την ενδιάμεση ε, αναθεώρηση και αν κοιτάξουμε την πορεία των εργασιών θα μπορούσαμε να πούμε από τη μία πλευρά έχει καταγραφεί πρόοδος, από την άλλη πλευρά υπάρχουν ορισμένες απώλειες και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ με αυτό. Ξεκίνησα τη χρονιά έχοντας στόχο να εδραιώσω τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα με απασχόλησε η κοινή η αρχή της κοινή δήλωσης. Ε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Μας επιτρέπει να συμφιλιώσουμε, να συγκεράσουμε τα συμφέροντα των περιβαλλοντικών ομάδων και τα συμφέροντα των μεταφορέων. στα ποτάμια και στα κανάλια. Τι, θα, τι κάνουμε λοιπόν με την κοινή δήλωση. Ζητάμε από από τους ενδιαφερόμενους ε, να επικοινωνήσουμε, να, δημιουργήσουμε μια συντονιστική ομάδα έτσι ώστε να βρίσκεται το θέμα στα χέρια όλων και να μπορούν να, να παρεμβαίνουν ανα πάσα στιγμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τώρα στο Δούναβι. Υπάρχουν δύο σχέδια που συμπεριλαμβάνουν την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Το ένα είναι μόνο η Ρουμανία, το άλλο είναι κοινό. Στη Ρουμανία τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ήταν ένα, ένα έργο της ΣΥΣΠΑ, τώρα ε, ανήκει στα διαρθρωτικά ταμεία και αυτό τους δίνει και περισσότερο χρόνο και περισσότερο χρήμα. Πολύ σημαντικό. Τι θα κάνουμε τις ε, δύο επόμενες, ε, τα δύο επόμενα τρίμηνα θα γίνει καταρχάς μια παρακολούθηση, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Και μετά θα ξεκινήσει η, ε, το έργο. Νομίζω ότι είναι καλά αυτά τα νέα θα παρακολουθήσουμε και τα όσα συμβαίνουν στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, μετά θα περάσουμε στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία γίνεται μία μελέτη, πήγε καλά η μελέτη. Στην ε, Ουγγαρία άλλαξε αρκετές φορές η κυβέρνηση. Κάτι που δυσκόλεψε τα πράγματα γιατί κάθε φορά χρειαζόταν να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Μια που κάθε υπουργό χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να εξοικειωθεί ναι, ένα καφέ θα τον ήθελα πάρα πολύ. δεν μου αρέσει να εργάζομαι σε μια χώρα που η κυβέρνηση δεν ξέρει ακόμα τι κάνει. Λοιπόν θα πρέπει να περιμένω να εξοικειωθεί η κυβέρνηση με τα πράγματα και μετά να συνεργαστούμε. Ουγγαρία και Σλοβακία βρίσκονται σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη θέση. Οι περισσότεροι θέλουν κάτι, αλλά δεν είναι πάντοτε το ίδιο αυτό που θέλουν. Να περάσω τώρα στην Αυστρία. Όταν αναφέρθηκα σε απώλειες, εννοούσα την Αυστρία. Στην αρχή η Αυστρία ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Υπήρχε ένα θαυμάσιο πρόγραμμα, ένα θαυμάσιο έργο στην υπέροχη αυτή χώρα με το υπέροχα τοπία ξαφνικά διαπιστώθηκε ότι η άδεια δεν ήταν σωστή και έχω την εντύπωση ότι θα φτάσουμε στο 2022 πριν να είναι έτοιμη είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να το συμπίσουμε. Περνάμε στα δύσκολα τώρα στην ε, Γερμανία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του Δούναβη γιατί εκεί ακριβώς ε, συναντάτε με το Ρήνο Υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών περιοχών. Ξεκίνησε λοιπόν μια μελέτη στο σημείο αυτό, όπου είπαμε ότι συναντώνται ο Μάιν, ο Ρήνος και ο Δούναβης, και έχουν συνυπολογιστεί όλες οι πτυχές, έχουν ακουστεί οι γνώμες όλων, των μεταφορέων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Επισήμως αναφέρεται ότι όλα βαίνουν καλώς. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε και αυτό. Το Σένα Νόρ δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα, τουλάχιστον προβλήματα που να βγαίνουν προς τα έξω. Εδώ όμως ένα οικονομικό που θα πρέπει να τεθεί. Πόσο θα είναι το τίμημα, πόσο ψηλά ε, θα φτάσουν τα διόδια. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή. Ελπίζω οι προσπάθειές μας να στεφτούν από επιτυχία γιατί το Σένενορ αφορά αρκετές περιοχές. Το Βέλγιο και η Ολλανδία ετοιμάζονται την ημέρα που θα ανοίξει η διόρυγα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή όταν Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάιλ. Θα προχωρήσουμε τώρα ε, στον κύριο Βαλέντε Ταριβιέρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ε, επαναλάβω το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκα πέρσι, διότι παραμένει το ίδιο. Οι δυνατότητες της Ευρώπης όσον αφορά τους λιμένες είναι μεγάλοι. έχω συνεχίσει τις διαβουλεύσεις μου με τους ε, Ευρωπαίους ενδιαφερομένους, τους stakeholders. Έχω συνομιλήσει με πάνω από 300 ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Έχω συναντηθεί με ναυτικούς, ε, με πλοηγούς, ε, έχω συνομιλήσει λοιπόν με πολλούς και σε έναν ε, μήνα θα έχω ολοκληρώσει τις συζητήσεις αυτές. Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα. Θα θυμάστε ότι υπήρχε σημαντική ανησυχία σχετικά με τις υποψηφιότητες. Μπορώ να σας πω ότι φέτος ε, έχει αντιστραφεί η τάση με βάση τις ε, συστάσεις από την προηγούμενη έκθεσή μου η Κομισιόν ε, με στήριξη των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να αλλάξει τις προτεραιότητες και να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασίας. Οι τροποποιήσεις αυτές αποδείχθηκαν πολύ θετικές μέχρι στιγμής. Έχουμε λάβει λοιπόν 14 επιλέξιμες προτάσεις που αντιπροσωπεύουν ε, συνολικές επενδύσεις σχεδόν 750 εκατομμυρίων ευρώ και Ε, ζητείτε χρηματοδότηση 185 εκατομμυρίων ευρώ πάνω από το διπλάσιο της, ε, των διαθέσιμων πόρων. Όσον αφορά λοιπόν ε, την εσωτερική αγορά, την, το παγκόσμιο εμπόριο, την ασφάλεια των πλοίων, τους λιμένες, ε, τις αλυσίδες τροφοδοσίας, σε προηγούμενες εκθέσεις έχω αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να τα εξετάσουμε όλα αυτά και στην έκθεση αυτή έχω προσθέσει δύο πράγματα. Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ανθρώπων που ε, ασχολούνται με τις μεταφορές και ε, αναθεώρηση των στρατηγικών κατευθύνσεων, διότι Υπάρχουν πολλές επιλογές και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας το εμπόριο με την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο, αλλά έχουμε την Κίνα, το, τη Σιγκαπούρη, το Σουέζ και τη Μεσόγειο σαν ε, σημαντικές περιοχές. Επιμένω λοιπόν στη σημασία του ανθρωπίνου στοιχείου στην αλυσίδα των μεταφορών. Ε, επιμένω λοιπόν στην ε, ε, επαγγελματική κατάρτιση. Θα σας αναφέρω τις 16 συστάσεις που έκανα, είναι πάρα πολλές, τις περισσότερες όμως τις γνωρίζετε από προηγούμενες εκθέσεις. Θα σας τις διαβάσω για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Προτείνω να εξεταστεί η ανάπτυξη ε, ολοκληρωμένης υποδομής για τους λιμένες ε, τα συστήματα πληροφορικής, ε, την κίνηση των εμπορευμάτων, τα οχήματα κλπ. Δεύτερον, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις πήγες υποδομές. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη. Μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι δρόμου, ένα μικρό κομμάτι σιδηρόδρομου. Κάποιο υδραγωγείο, μερικές φορές μπορεί να μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις ε, επίγειες συνδέσεις, θα πρέπει να ε, εξετάσουμε τους, ε, τους κρίκους της αλυσίδας που απουσιάζουν. Κινητοποίηση ε, εφιών υπηρεσιών υποδομής. Να βελτιώσουμε την ασφάλεια και να ε, επιτρέψουμε τον πλήρη έλεγχο ε, συστημάτων τα οποία να παραδίδονται και εγκαίρως. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, μια υπηρεσία ασφάλειας ε, που εδρεύει στην Λισαβόνα, η ΕΜΣΑ, και προτείνω να την επισκεφτείτε, διότι είναι πολύ καλή ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία ε, ήδη κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι διατεθειμένη να κάνει ακόμα περισσότερα. Η τέταρτη σύσταση είναι να προωθήσουμε δραστηριότητες και μελέτες για να καταλάβουμε καλύτερα τον ε, τομέα αυτών. Επιμένω, οι ε, μελέτες είναι απαραίτητες ε, για να καθορίσουμε τη δράση μας. Θα πρέπει να εξετάσουμε τους, τις δραστηριότητες των λιμένων. Πολλά μέρη της Ευρώπης θέλουν να αποτελούν κόμβο και είμαι υπέρ αυτού διότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα μεγάλα κέντρα μεταφορών, τους κόμβους δηλαδή. Η Ευρώπη με τόσο μεγάλο μήκος ακτών πάνω από 95.000 χιλιόμετρα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε κομβικά σημεία με ακτίνες ε, σχεδόν παντού και να αποφύγουμε τις οδικές μεταφορές και να τις ε, υποκαταστήσουμε με θαλάσσιες μεταφορές. Έκτον, Ε, οι ε, θαλάσσιες μεταφορές ε, θα επωφεληθούν πολύ από την βελτιωμένη κατάρτιση. Έχω προτείνει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Εράσμους για αυτό. Από ό,τι φαίνεται μόνο τρεις χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν πρόβλημα με την κατάρτιση του ναυτιλιακού προσωπικού. Όλες οι άλλες χώρες έχουν πρόβλημα και μπορούν να επωφεληθούν από το δίκτυο αυτό, εάν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί. Η έβδομη σύσταση είναι να αναπτύξουμε δράσεις και σύστημα πληροφόρησης ε, για να ε, έχουμε διαδικασίες ε, ενιαίας θηρίδας, one-stop shop. Υπάρχουν αρκετά καλά παραδείγματα αυτού και έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολύ χρόνο κατά τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να γενικευθεί το σύστημα αυτό και να υιοθετηθούν οι ίδιες διαδικασίες στο σύνολο της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη ε, τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο. Η έρευνα και η ανάπτυξη για να ε, αναπτυχθούν πλοία και εξοπλισμός που μειώνουν το, τις εκπομπές και αυξάνουν την ε, ασφάλεια και είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Έχω προτείνει να υπάρχει ε, όριο στην ηλικία των πλοίων και να βελτιωθεί η ποιότητά τους. Δεν θα κάνω πολλές άλλες προτάσεις ε, για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά να έχουμε κατά νου την απόδοση των πλοίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε επίσης ε, να είναι σαφή τα χρηματοδοτικά πλαίσια. Ήδη, και το είπα αυτό πέρσι, έχουμε ε, ένα χρηματοδοτικό μέσο για το ΜΟΣ. Ε, έχουμε όμως και Ταμείο Σύγκλησης, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το... Ο κόσμος χρειάζεται συμβουλές και πληροφόρηση σχετικά με τα ταμεία αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια υπηρεσία για ε, τη χρηματοδότηση και αυτό είναι πολύ θετικό. Προτείνω να ε, επικαιροποιηθούν οι κατευθυντήρες γραμμές ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τέντη και θα ήθελα να έχουμε κάτι αντίστοιχο με αυτοκινητόδρομους ε, στη θάλασσα ε, στα πλαίσια της τροποποίησης ε, των κατευθυντηρίων γραμμών αυτών. Απλοποιημένη γραφειοκρατία όπου αυτό είναι δυνατόν, βελτιωμένη λύση κάποιων ευέλτιστων πρακτικών και σας προτείνω να στηρίξετε το σύστημα Eurobonus. Οι Ιταλοί έχουν ένα σύστημα Ecobonus, οικολογικού πριμ και Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για την Ευρώπη να έχει ένα γενικευμένο σύστημα. Και γι' αυτό εγώ δεν το ονομάζω eco-bonus, το ονομάζω euro-bonus. Ε, αυτό δίδεται απευθείας στους οδηγούς. Και έτσι αποφεύγουμε ε, την... Ε, την ε, αυξημένη πίεση στους δρόμους, στις οδικές μεταφορές. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα το ε, εκομπόνους της Ιταλίας, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά υπάρχει ε, σημαντικός όγκος προβλημάτων με τους γειτόνους μας. Ε, και σε ποιους γειτόνους αναφέρομαι. Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, την Βόρεια Αφρική. Ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά ούτως ή άλλως είναι πολύ κοντά για να τους ξεχάσουμε, ε, για να τους παραβλέψουμε. Και έχουμε και, τους, έχουμε και τα ανατολικά μας σύνορα και εδώ έχουμε σημαντικά προβλήματα. υπάρχουν πολλά συμφέροντα από την άλλη μεριά και Δεν μπορούμε να του αρνηθούμε οποιαδήποτε στήριξη, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο. Θα πρέπει να εξετάσουμε τους λιμένες, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν διαφορετικό σύστημα. Το ρωσικό σύστημα είναι διαφορετικό από ε, το ευρωπαϊκό. Και θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Υπάρχουν και διαφορετικά είδη καυσίμων. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, διότι είναι πολύ πιο ασφαλές όσον αφορά τις ε, εκπομπές ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα, σωματιδίων κλπ. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο απαιτεί δίκτυο σημείων τροφοδοσίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα δίκτυο με σημεία τροφοδοσίας πολύ πιο κοντά από ό,τι ε, είναι αυτή τη στιγμή. Ε, όπως και να έχει όμως είναι πολύ πιο ασφαλές και πιο καθαρό από το παρόν σύστημα. Ήδη έχω αναφερθεί στην ανάγκη... Ναι, ναι, κλείνω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια πολιτική έρευνα για τις μεταφορές με σαφείς ε, τομείς προτεραιότητας. Κλείνοντας, ε, να πω ότι περιμένω ε, να υλοποιηθούν οι συστάσεις αυτές, οι οποίες έχουν εκπανηθεί κατόπιν συνομιλιών με Ευρωπαίους ενδιαφερομένους. Θέλουμε να πετύχουμε έτσι ε, βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχω τέσσερις συντονιστές και τρεις άλλους βουλευτές ε, στην δόση αυτή, να το πούμε έτσι. Οχτώ ομιλητές. Θα ήθελα να σας περιορίσω στα τέσσερα λεπτά τον καθένα, ώστε... να ακούσουμε τις απαντήσεις των συντονιστών. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων θα είμαι αυστηρός, όμως πρέπει να είμαι αυστηρός ε, για να προλάβετε να πάρετε όλο το λόγο. Ο κύριος Γκρός από τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συντονιστές, την Κάρλα και τον συνάδελφό της. Πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ε, γι' αυτό θα περιοριστώ και εγώ σε μερικά σημεία. Πρώτον, οι εκθέσεις από χρόνο σε χρόνο εμφανίζουν τις ίδιες καθυστερήσεις. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν ήταν πιο αυστηρή λίγο στις καθυστερήσεις στις συντονιστές γιατί η δική σας αποψή θα μας βοηθήσει να κάνουμε την αξιολόγηση και την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, με τρόπο έτσι πιο συγκροτημένο και πιο τεκμηριωμένο. Διότι Διαβάζω στην έκθεση της Κάρλα Πέις κάτι από μια χώρα που γνωρίζω καλά εγώ και το, ε, τις κάτω χώρες υπάρχουν συνεχώς συγκρούσεις ε, ε, για θέματα υποδομών και θέματα περιβάλλοντος. Ε, κάποιες προτεραιότητες δεν θα πρέπει επιτόπου να διεκπεραιώνονται πολύ πιο γρήγορα και να ορίζονται αντίστοιχα για να αποφεύγονται τέτοιες συγκρούσεις. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τη χρηματοδότηση. Το πρώτο, άκουσα κάτι για ε, σύστημα διοδίων ε, στη Γαλλία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με αυτό, ούτε ενισχώ ιδιαίτερα, αλλά μπορείτε να με ενημερώσετε τι λέει η έκθεση, πώς το φαντάζεστε αυτό, πώς θα ενσωματωθεί στην Ευρώπη. Και ένα δεύτερο υποερώτημα, κάτι που είπα και εισαγωγικά, η χρήση των χρημάτων στους δικούς σας τομείς, πώς γίνεται αλλά και στη δεύτερη έκθεση. Γιατί νομίζω ότι και αυτό κάπως ε, χρονοτριβεί από τα 85 εκατομμύρια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών, τα 60 πάνε στο Μάρκο Πόλο. Ε, πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια και ε, με ποια ταχύτητα και για ποιο σκοπό. Και μια τελευταία παρατήρηση. Κάνατε προτάσεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 12 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σας. Σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται και αντιστοιχούν στην πολιτική που επιθυμούμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να βρούμε όμως από κοινό δρόμο να πείσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και σε κάποιους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης να επενδύουν πολύ περισσότερο για να έχουμε και λιμένες και καλύτερη σύνδεση και διασύνδεση με την χώρα. και είναι και ε, κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς να έχουμε πιο συγκροτημένη συζήτηση με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα για μας, πώς μπορούμε καλύτερα να συντονιστούμε και με μεγαλύτερη συνοχή πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό έρχεται εδώ να είναι ε, να γίνει ενδιαφέρουσα η δική σας έκθεση και για τη δική μας Επιτροπή για την ενδιάμεση αναθεώρηση και τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Θα πρέπει όμως να έχουμε μια σαφή πολιτική, συγκεκριμένη και συνεκτική. Παρακαλώ, πείτε τα αυτά και στον Επίτροπο που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος. Διότι εδώ μας λείπει η συνοχή και θα πρέπει περισσότερο να μας βοηθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλχαντράουι από τους Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντονιστές των δικτύων για την καλή δουλειά τους και την καλή εισαγωγή τους. Κυρία Πέις, θα ήθελα καταρχάς να σας πω για το Δούναβι ότι η κυρία Τσικάου που είναι πολύ ειδική στο Δούνα, δυστυχώ σήμερα ε, και δεν παρευρίσκεται. Δεν θα μακρηγορήσω εγώ για το Δούναβι, αλλά και πάλι βλέπουμε καθυστερήσεις και ε, που συνδέονται με αλλαγές κυβερνήσεων. Έρχονται και παρέρχονται κυβερνήσεις και η δική σας εμπειρία τι λέει, μπορείτε να κάνετε συστάσεις για το μέλλον. Πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πώς βλέπετε το ρόλο των συντονιστών, ίσως ένα πιο ισχυρό ρόλο για τους συντονιστές για να ε, μην έχουμε τέτοιες χρονοτριβές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχει πιο ισχυρή παρουσία. Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Σικουάνα με τη Βόρεια Θάλασσα, τη διόρυγα Σεν Νόρ, από ό,τι φαίνεται ε, ε, είναι οικονομικό το πρόβλημα και άκουσα κάτι για σύστημα διοδίων. Και ποιο θα ορίσει το ύψος. Πόσο θα είναι αυτά. Ε, θα είναι κάτι σαν το BPS. Κάτι άλλο που διαβάζουμε και στην ενδιάμεση αναθεώρηση είναι ότι κινδυνεύει να μειωθεί η συμμετοχή ε, στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή όταν είναι ιδιαίτερα μεγάλες οι καθυστερήσεις, να παίρνονται πίσω τα χρήματα και να πηγαίνουν σε άλλα έργα. 44,3 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή ευρωπαϊκά κινδυνεύουν να ε, στραφούν αλλού. Και τέλος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε γρήγορα θα πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε ε, με τη φάση της μελέτης, να μπει και καμιά μπουλντόζα να αρχίζει να σκάβει τώρα εκεί στα έργα. Εντάξει μελέτες. Και για τον κύριο Βαλέντε Ντολιβέρα θα ήθελα ε, να πω το εξής. Διάβασα το σημείωμα και αυτό που συγκρατώ είναι ότι δεν ενδιαφέρεται ο κλάδος ε, να προχωρήσει βλέπω ανέβετε κι εσείς και συμφωνείτε σε αυτό, αλλά μπορείτε να μας δώσετε καμία ένδειξη <laughs> για το πώς θα έχουμε πρόοδο σε αυτό το τομέα. Και τι σας απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες αυτές τις στάσεις που σας απευθύνεται μελέτες, benchmarking, συγκριτική αξιολόγηση έχει αντιδράσει με κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αντιδράσει, πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάισνερ από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, δεν χρειάζεται να μιλήσω για τέσσερα λεπτά. Έχω μία ερώτηση ε, προ την κυρία Πάη. ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομα, γιατί είναι στρατηγική του Δουναβή. Κατάλαβα σωστά ότι ε, έχει ξεκινήσει η παρακολούθηση ε, των Κυπρίνων στην περιοχή, διότι αυτό είναι ένα ψάρι. Α, και επίσης όσον αφορά Ε, Τη μεταφορά λέμε ότι είναι πολύ πιο ε, οικολογικέ οι θαλάσσιες μεταφορέ από ότι οι οδικέ. Ε, έχω μιλήσει στη Γερμανία με το σχετικό κλάδο και μου ανέφεραν τεράστια ποσά όσον αφορά τι δυνατότητε των θαλασσίων μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και ε, οικολογικά τι θα ήταν σκόπιμο κατά τη γνώμη σας. Και ε, άλλη ερώτηση. Ε, αναφέρατε τις καλύτερες αλυσίδες τροβοδοσίας υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ε, ίσως αυτό αφορά και τους δύο μιλητές. Τέταρτη ερώτηση. Μιλήσατε για πιο πράσινη ναυτιλία, κύριε Ολιβέηρα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να ρωτήσω όσον αφορά τις δυνατότητες της Ευρώπης, τι θα ήταν απαραίτητο για να πετύχουμε μείωση των εκπομπών των πλοίων. Και ε, ο κύριο Ολιβέηρα μίλησε και για μείωση τη γραφειοκρατία. Φυσικά αυτό το θέλουμε όλοι. Έχετε ε, συγκεκριμένα παραδείγματα, ε, διότι άλλο το να μιλάει κανείς θεωρία, άλλο το να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με τα οποία να μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Λίχτεμπεργκερ ε, για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τις ε, ομιλίες που ακούσαμε. Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα όσα άκουσα από τον κύριο Βαλέντε Ντολβιέρα το ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος ε, στο θέμα της, ε, των θεμάτων της αλυσίδας ε, τροφοδοσίας. Πιστεύω ότι είναι σωστή η προσέγγιση αυτή. Εάν δεν μπορούμε να φέρουμε τα αγαθά στο λιμένα, τότε δεν έχει πολύ νόημα να έχουμε εκεί σημαντικές υποδομές. Ε, και θα ε, αναφερθώ πολύ σύντομα στο θέμα του Δούναβη. Επισκεφτήκαμε τον Δούναβη και είδαμε ότι το δυναμικό αυτή τη στιγμή δεν εξαντλείται διότι ε, διότι έχουμε πολύ μεγάλο όγκο προβλημάτων όσον αφορά τους χώρους μεταφόρτωσης, ε, την ε, την μεταφορά των αγαθών και τα λοιπά. Και αυτό είναι αποφασιστική σημασία για μένα. Ε, εμένα δεν με στεναχωρεί Ε, τόσο που δεν, ε, θα γίνει, που δεν θα γίνει εξκαφή ακόμα στο αυστριακό κομμάτι. Ε, ίσως ε, καταλήξουμε να προσαρμόσουμε τα πλοία στο ποτάμι. Ε, ερώτησή μου. το πρόβλημα του Δούναβη θα ε, συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και εάν γίνουν οι εξκαφές. μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μπορούμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, διότι εγώ βλέπω τη δυνατότητα αύξησης του δυναμικού στο Δούναβι, κυρίως στον τομέα αυτών, με την βελτίωση δηλαδή της, ε, των αλυσίδων τροφοδοσίας ε, και με προσαρμογή των πλοίων στο ποτάμι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο οικολογικό. εάν το 80% των, εσωτερικών, των ναυτιλιακών μεταφορών εσωτερικών υδάτων ε, γίνεται στο Δούναβι, τότε θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη στην ε, όλη ε, προοπτική. Και θα πρέπει η προσέγγιση μας να προσανατολίζεται περισσότερο στο θέμα της τροφοδοσίας, της επιμελητίας και Θα μπορέσουμε έτσι να πετύχουμε ε, πρόοδο στο θέμα της μεταφοράς αγαθών. Ε, πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάποιες ε, διαμάχες. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε λύσεις όμως που να μην μας οδηγήσουν σε αναμονή 5, 10, 15 ετών μέχρι να εξαντληθεί το δυναμικό του Δούναβη και θα ήθελα να προτείνω μία συντονισμένη μελέτη ε, για το σύνολο του Δούναβη. Τι αγαθά μεταφέρονται στο, ε, στην περιοχή αυτή και τι προβλέπετε όσον αφορά τις ε, ανάγκες για δυναμικό στο μέλλον. Ευχαριστώ. ακούσαμε τους ε, των πολιτικών ομάδων. Τώρα προχωράμε στους μεμονωμένους ομιλητές. Παρακαλώ. Πιστεύω ότι οι δρόμοι της θάλασσας είναι δύο σημαντικοί άξονες που θα πρέπει να έχουν όλη μας τη στήριξη. Η κυρία Πέις μίλησε εδώ για το Δούναβι, διάβασα βεβαίως την έκθεσή της. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αυτή είναι μία ευχή. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες λεωφόρους, κοιτάζοντας προς Ανατολάς, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να κοιτάξουμε προς την Αδιατρική και μετά προς ε, την Τρινική θάλασσα σε μία προσπάθεια να αναπτύξουμε το εσωτερικό της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε φορείς μια σημαντική δύναμη στον τομέα της, ε, των μεταφορών. Βεβαίως ε, γι' αυτό απαιτείται μια σωστή διάρθρωση στα λιμάνια και στις άλλες μετα, μεταφορές των, ε, υποδομές των μεταφορών. Θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τις μεταφορές στις πλωτές οδούς. Ευχαριστώ κύριε Ολιβέρα που αναφερθήκατε σε αυτή την δυνατότητα του Ιταλικού εκοβόνους Πιστεύω ότι μια ευχή είναι να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό αερομέονους. Δεν θέλω να σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Εσείς που ασχολείστε με αυτά τα θέματα, επειδή έχετε εντοπίσει το θέμα του προγραμματισμού, τα προβλήματα που βρίσκεται αφορούν τις διαδικασίες, τη γραφειοκρατία, το κόστος. Την ερώτηση αυτή την κάνω για να καταλήξω στο εξή. Όταν εντοπίσατε αυτά τα προβλήματα, ποια είναι η δική σας ανάγκη για να μειώσετε το χρόνο, για να επιτύχετε περισσότερα αποτελέσματα, για να έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε όσο γίνεται πιο σύντομα αυτό το θέμα ή το πέρασμα από τις οδικές μεταφορές στις θαλάσσιες μεταφορές. Ποια είναι η δική σας άποψη, ποιο είναι το δικό σας συγκεκριμένο αίτημα έτσι ώστε όλα αυτά να μπορέσουν να γίνουν πιο επικοδομητικά όσο γίνεται πιο σύντομα. Πέρα βέβαια από το θέμα των οικονομικών που θα πρέπει να το συζητήσουμε ε, σε ένα επιμέρους κεφάλαιο. Ο κύριος Σέζου. Ευχαριστώ. Ε, έχω μερικά σημεία να σας ε, θέσω υπόψη, κυρία Πέης, και σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Εγώ είμαι από την κάτω Βαβαρία, σοσιαλδημοκράτης και έχω διαδεχθεί τον κύριο Γκέρχαρτ Σμιτ, ο οποίος σας στέλνει και τους ε, φιλικούς του χαιρετισμού. Θα ήθελα να σας πω μερικά σημεία να λάβετε υπόψη σας τις αποφάσεις που θα λάβετε για τα έργα εκεί. Πρώτον, μιλήσατε για την ομάδα παρακολούθησης και ελέγχου του 2008, ε, Monitoring Group, και ε, την αντίστοιχη μελέτη που έχει ανατεθεί, η οποία είναι καθοδόν ακόμα. Γνωρίζετε ε, ε, ότι έχει ανατεθεί στην RMD Wassenstrasse GmbH απευθεία ανάθεση, θα το γνωρίζετε ε, μια εταιρεία που το πήρε με άμεση ανάθεση θηγατρική της RMD που είναι Rhinos Main Donau και το πήρε χωρίς διαγωνισμό χωρίς κανέναν ανταγωνισμό με απευθείας ανάθεση και αυτοί όλοι εντάσσονται στον ε, όμιλο αίων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όποιος ξέρει ε, τι είναι η εταιρεία αίων που παράγει ε, ενέργεια και θέλει να συμμετέχει σε αυτά τα έργα. Δεύτερον, η Γερμανία σύμφωνα με το άρθρο 326 ε, υπέρ μιας έρευνας αντικειμενικής και ανεξάρτητης και είναι ε, αρμόδια Γερμανία και ο Υπουργός Ραμζάουερ ε, έχει ζητήσει την επιλογή του σε 280 27 Ιουλίου ε, η Πάσα ΕΠΡΕΣΕ, η τοπική εφημερίδα τα αναφέρει αυτά τα πράγματα. Ο Υπουργό δεν έχει το δικαίωμα να υποδεικνύει τι θέλει. Η ομάδα παρακολούθηση λοιπόν στελεχώνεται από ειδικού τη εταιρεία αυτή, τη RMD, και ε, μάλλον όχι, έχει συμβούλου αυτή τη εταιρεία και έχει συμβούλου του Υπουργείου. Πώ γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι δυνατά. Σα παρακαλώ κυρία Πέη, όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη σα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, και προτεραιότητα για τη δική μου περιφέρεια. Και δεν θέλουμε και στην, νότια Βαβαρία, στην κάτω Βαβαρία συγγνώμη, ένα έργο τύπου Στουτκάρδη 21 που έχετε δει τι χαμός γίνεται εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Εζόκ. Αγαπητά μέλη, ο κατάλογος γίνεται όλο και πιο μακρύς από τα ονόματα που προστίθενται. Αν συνεχίζετε λοιπόν Λοιπόν, να προσθέτετε ονόματα θα χρειαστεί να μειώσω το χρόνο αγόρευσης. Κυρία Βιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Πέις και τον κύριο Βαλέντε Ε, θέλω ερώτηση να κάνω στον κύριο Βαλέντε. Ενδιαφέρονται αυτά που μας είπατε. Αλλά κάτι που μου λείπει από όλη αυτή την προσπάθεια είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωραία, οι αναλύσεις είναι καλές. Συμφωνούμε όλοι ε, γενικά ε, για τις συστάσεις σας. Οι συστάσεις... ε, είναι κάτι στο οποίο δίδεται συνέχεια και θα δείτε στο μέλλον. Αλλά αυτό που μου λείπει είναι μεγαλύτερη ακρίβεια, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα. Για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα ευρωπαϊκό έργο, συνολικό όμω, όπου στι συστάσει να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και κάποιε πρωτοβουλίε που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα και να δούμε πώ μπορούμε σιγά σιγά να οικοδομούμε το μέλλον. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα εγκρίναμε τους σιδηροδρομικούς διαδρόμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα επιθυμούσα οι συστάσεις που μιλάει και για τις διασυνδέσεις ε, των σιδηροδρόμων με τις λεωφόρους της θάλασσας. Να, να τα δει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τα εξετάσει αν είναι καλό το έργο, πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να προωθηθεί. Αυτό ακριβώς μου λείπει στις συστάσεις πολύ θεωρητικές είναι και ασαφείς και αόριστες. Δεν θα πρέπει αυτά να τα συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια στιγμή. Τα έργα που ήδη γίνονται να κάνουμε μια αξιολόγηση αν είναι εύστοχα προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, εσείς μιλήσατε για τα έργα που υπερβαίνουν σε κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ ε, τα κονδύλια που διαθέτουμε και σας ερωτώ τώρα με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν τα διάφορα έργα αν δεν φτάνουν τα χρήματα και αν υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλογής μεταξύ αυτών θα λαμβάνονται ε, υπόψη ε, τα έργα που ήδη τρέχουν, η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, της εσωτερικής αγοράς. Και όταν μιλάτε για ανάγκη ε, εξυγχρονισμού των μεταφορών μέσω επενδύσεων και καινοτομίας, έχετε λάβει υπόψη σας και τα ναυπηγεία στην Ευρώπη. Είναι στρατηγικός τομέας. Πρόσφατα το εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη σύνοδο στο Στρασβούργο. Η θάλασσα λοιπόν είναι στρατηγικός τομέας και ε, η ναυπηγική ε, βιομηχανία περνάει πάρα πολύ ε, δύσκολες στιγμές από τον ανταγωνισμό της Νοτιοανατολικής Ασίας. Καλή ενιαία θηρίδα, ωραία όλα αυτά που λέτε και είναι ένα στοιχείο που θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό έργο σχέδιο. Θα σας υποστηρίξω πλήρως εκεί, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία, διότι θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη. Όλοι μαζί θα πρέπει λοιπόν να οικοδομούμε ευρωπαϊκά επαναλαμβάνω έργα και όχι εθνικά έργα. Γιατί έχουν αντιστάσεις τα κράτη και θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε αυτό και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε όλη μου την υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή για να μιλήσετε για τις θαλάσσιες λεωφόρους. Θα ήθελα κυρίως να σας συγχαρώ για την προσοχή που δώσατε για, τις, για περιοχές όπως η Μαδέρα από όπου προέρχομαι που έχει <clears throat> εδαφικές ιδιαιτερότητες που δεν λαμβάνονται συχνά υπόψη. Η μεταφορά αγαθών στην περιοχή, στις περιοχές αυτές είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία και το εμπόριο. Είναι και για τον τουρισμό και για την κοινωτικότητα των ατόμων. Το 5% των προϊόντων που καταναλώνται στη Ματέρα είναι εισαγόμενα. Και τα περισσότερα από αυτά έρχονται με θαλάσσιες οδού. Γι' αυτό το λόγο οι θαλάσσιες μεταφορές είναι τόσο σημαντικές, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά όπως πολύ σωστά λέτε κύριε καθηγητά στην έκθεσή σας, παίζει ρόλο και η στρατηγική θέση αυτών των περιφερειών. Στην πολιτική έκθεση ενεκρίθη μία, μία τροπολογία στην οποία αναφέρεται ότι η Ένωση έχει την καλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη γιατί υπάρχουν αυτές οι, ε, οι, απομακρυσμένες περιφέρειες. Αυτή είναι μία άποψη που συμμερίζομαι. Οποιαδήποτε οτιδήποτε αναγνωρίζει αυτή την ιδιαιτερότητα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της Επιτροπής για την εφαρμογή αυτών των μελετών που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κυρίως τις θαλάσσιες λεωφόρους στις απομακρυσμένες περιοχές. Ποια είναι, ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, πόσο ανοιχτή είναι η Επιτροπή για τέτοια προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένη. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Ολιβιέρα είναι... σχετική με το θέμα ότι στην ενδιάμεση αναθεώρηση δεν μπορούσα να βρω κανένα στοιχείο σχετικά με ε, το έργο υπαριθμών 21. Ε, είναι ένα σύστημα που αφορά τη Βαλτική. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό, διότι βλέπω να υπάρχει η δυνατότητα εδώ να ε, συνενώσουμε δύο προγράμματα, το 21 και το 27. Και έτσι μπορεί να φέρνει κανείς τα εμπορεύματα μέσω των λιμένων και κατόπιν να ε, μεταφορτώνεται στους ε, σιδηροδρόμους. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τις ε, εκπομπές του άνθρακα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι θα γίνει με τα δύο προγράμματα αυτά στο μέλλον. Ίσως είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου, αλλά ε, είμαστε πολύ συναδελφοί από τις χώρες του Βορρά και της Βαλτικής. Οπότε Ευχαριστώ. κύριο ε, ε, ο κύριος Κράμερ, ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ έχω μια ερώτηση σχετικά με την ναυτιλία εσωτερικών υδάτων. Το 80% πραγματοποιείται στον Ρήνο, λέγεται, και αυτό είναι πολύ καλό. Στον Δούναβη θέλουμε να δημιουργήσουμε συμφόρηση. Μου φαίνεται εμένα ότι το λόμπι των κατασκευών βρίσκεται από πίσω. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι. Εγώ από το Ingolstadt μέχρι την ε, ε, ε, Μαύρη Θάλασσα έχω στο Δούναβη και είναι πλωτός ο Δούναβης ε, για τα τρία ή τέσσερα αυτά μεγάλα πλοία που θέλουν να πάνε από τον Ατλαντικό στην ε, Μαύρη Θάλασσα ε, θα κάνουμε τέτοια έργα. Μπορείτε οικονομικά να μου αιτιολογήσετε γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Στα μεγάλα προγράμματα η σχηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 25% για τους δρόμους της Βαλτικής για παράδειγμα είναι 10% επειδή μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα αυτό το επιχείρημα, το σωστό επιχείρημα δεν το έχω ακούσει ε, ακόμα. Ε, η ερώτησή μου είναι λοιπόν πόσα πλοία υπολογίζεται να υπάρχουν. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μείωση από 20 σε 8%. Ε, γιατί ε, καθυστερείται πήγοντα έργα εάν δεν λάβουμε απάντηση σε αυτό δεν θα μπορέσω να πείσω κανέναν ούτε στο Χάινμπουργκ, ούτε στο Δούναβι, ε, ούτε στη Γερμανία, ούτε πουθενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Βαλέντε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που έθιξε ο συνάδελφος Τεξέρα, όχι για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιοχές, αλλά για, τις, ε, για τα νησιά της Μεσογείου. Στις συστάσεις δεν άκουσα να γίνεται καμία αναφορά στην έκθεση που υπάρχει μεταξύ της, ε, του νησιώτικου χαρακτήρα των περιοχών και των θαλασσίων λεωφόρων. Θα ήθελα να κάνω αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Στις ε, διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν, βρήκατε στοιχεία για να επανεξεταστεί η πολιτική για το υποχρεωτικό καμποτάζ. Δεύτερον, είναι δυνατόν μεταξύ των συστάσεων που θα κάνετε στο μέλλον να απαιτηθεί η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της διευκόλυσης των ε, συνδέσεων με τις νησιώτικες περιοχές. Τρίτον, εάν είναι προς επανεξέταση το κριτήριο που απέκλειε τη μεικτή σχέση ατόμων και εμπορευμάτων. Δηλαδή, ε, διευκολυνόταν η διακίνηση των αγαθών χωρίς αυτό να φύγει τη σχέση μεταξύ ε, ε, αγαθών και προσώπων. Ευχαριστώ. Η Αγιάλα Σέντερ, τελευταία για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω τους δύο εισηγητέ μας για λόγους κυκλοφοριακής συμφόρησης στην είσοδο των Βρυξελών. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στον κύριο Βαλέντε Ντε Ολιβέιρα σε σχέση με τις θαλάσσιες λεωφόρους και τα hubs που ε, προσπαθούμε ε, αυτοί οι κόμβοι να είναι ηλιμένες στα επόμενα δίκτυα, να ανακτήσουν αυτό το ρόλο που δεν ποτέ έπρεπε να είχαν χάσει έτσι κι τα λιμάνια, στα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα. Μας έχετε δώσει κάποια στοιχεία. Ο βοράς ε, έχει το 75% του φόρτου και τα νότια λιμάνια είναι περίπου καταρχήν στο 25% του, του φορτίου του μεταφερόμενου. Και Λέτε ίσως ότι το πρόβλημα του Νότου είναι η πληθώρα λιμένων. Και η λύση ποια θα ήταν. Να έχουμε κλάστερ, να συνενωθούν τα διάφορα λιμάνια ή ε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Η έλλειψη ε, διασύνδεσης, ε, διαλειτουργικότητας με αυτοκινητοδρόμους, με σιδηροδρόμους ή έλλειψη σύνδεσης με την ενδοχώρα και άλλα στοιχεία. Φταίει μόνο το γεγονός ότι είναι πολλά τα λιμάνια. Η λειτουργία τους ίσως μήπως δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικά υπό την έννοια της απελευθέρωσης ε, των υπηρεσιών ή έλλειψη προσωπικού. Εσείς επανειλημμένα μας λέτε ότι χρειάζεται καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό. Ε, θα μπορούσατε να το εμβαθύνετε αυτό λίγο. Ε, πολλές φορές αναφέρατε την έλλειψη του ενδιαφέροντος του κλάδου για τα έργα αυτά των θαλασσίων λεωφόρων. Εμείς πιέζουμε τον κλάδο αλλά φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν. Και στο Μάρκο Πόλο καμιά φορά, συχνά μάλιστα, βλέπουμε ότι δεν ενδιαφέρονται. Ε, εσείς το έχετε αναλύσει αυτό, όλα τα έργα που έχουν κατατεθεί και στη Μεσόγειο. Έχετε συζητήσει και με τους πελάτες. Τι λέει αυτός ο κλάδος. Ποια είναι η ζήτηση στο κάτω-κάτω. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν θαλάσσιες λεωφόροι, κυρίως στη Μεσόγειο, που δουλεύουν ρολόι και υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση. Το έχετε κοιτάξει αυτό, το έχετε μελετήσει. Ή μήπω προτείνουμε ε, ε, στους ενδιαφερομένους στην οικονομία, στον κλάδο, έργα που δεν τους ενδιαφέρουν. Ε, τους προτείνουμε πράγματα που να θέλουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που πειθαρχήσατε. Ευχαριστώ κυρίως την κυρία Ντουράνη που αφαίρεσε το όνομά της από τον κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 15 λεπτά στη διάθεσή μας για να δώσουμε το λόγο στους εισηγητές. Με θερμινευόμενο σημαίνει 15, 17,5 ε, λεπτά ανά εισηγητή. Ωραία λοιπόν, κάντε μια προσπάθεια να ε, περιοριστείτε σε αυτά τα 7,5 λεπτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Και αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω Ολλανδικά. Για τον κύριο Γκρός. συνολική προσέγγιση με τη στρατηγική για το Δούναβι είναι δεδομένη αυτή και εξασφαλισμένη. Τι τέσσερις συντονιστές πήγαμε και θα, πάμε μάλλον σε λίγες εβδομάδες στην Ουγγαρία για να δούμε ε, πώς θα συνεργαστούμε οι βιομηχανικές περιφέρειες, ας πούμε, οι αυτοκινητόδρομοι, οι σιδηρόδρομοι και ο Δούναβης, για να μην έχουμε επικαλύψεις και επαναλήψεις. Θα το συζητήσουμε αυτό στην Ουγγαρία. Ευθύ εξ αρχής θεωρούσαμε το Δούναβη όχι μόνο πλωτίοδο μεταφοράς, αλλά και ε, ως οικοσύστημα. Ξέρετε, ο Δούναβης είναι ένα ποτάμι που ε, υπερχιλίζει και είναι ένα οικοσύστημα. Λοιπόν, κοιτάξαμε όλα αυτά τα θέματα, το πόσιμο νερό, τα πάντα να βεβαιωθούμε ε, και παραγωγή ενέργειας στη Σλοβακία. Δεν είναι μόνο η ναυσιπλοεία που μας ενδιαφέρει να περνάνε τα πλοία από το Δούναβι, αλλά και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Αυτά τα ξέρουμε και προσπαθούμε να ε, έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στο ποτάμι αυτό, η οποία έρχεται να ενισχυθεί από τη στρατηγική για το Δούναβι που δημοσιεύθηκε πλέον. Δεν είμαστε δηλαδή προσκολλημένοι στο, στον ποταμό, αλλά και τις γύρω περιφέρειες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και ξέρετε ότι είναι και διεθνές ποτάμι, περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Περίπου είναι οι κινέζικες διαστάσεις αυτές και μεγέθη. 3.000 χιλιόμετρα δούνευης ε, περίπου και ε, το λαμβάνουμε υπόψη. Ε, βεβαίως θα πρέπει να γίνει απαραίτητη ε, υποδομή. Κανένας δεν πρόκειται, και το λέω και στον κύριο Κράμερ, να επενδύσει εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ε, αριθμός ε, ημερών ε, που να είναι εγγυημένη η ναυσιπλοεία για συγκεκριμένα πλοία. Ας πούμε από 300 μέρες είναι πλωτός ο Δούναβης το χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τα μεγάλα καράβια. Και εγώ όταν είμαι στο δούναβη, βλέπω τέσσερα πλοία τη μέρα να περνούν. Ενώ ε, χρειάζεται ε, ε, πολύ μεγάλη προσοχή και καλός σχεδιασμός. Και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται με οικολογικό και καθαρό τρόπο. Να είναι καθαρά και τα πλοία και να ε, χρειαζόμαστε εκεί ερευνητικά κονδύλια γιατί υπάρχει πρόβλημα με τους κινητήρες των πλοίων. Είναι πολύ μικρή αγορά. Όταν κάποιος κατασκευάζει ε, ε, κινητήρες για πλοία δεν έχει τεράστια αγορά. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Και θέλω να ζητήσω και από το Κοινοβούλιο να το κοιτάξει αυτό. Γιατί καμιά φορά έχουμε ε, τους ίδιους ε, κινητήρες στα πλοία της εσωτερικής ναυσιπλοείας, κινητήρες που βλέπουμε που βλέπουμε σε μηχανήματα. Το πρόβλημα είναι το, το βαρύ πετρέλαιο, δεν είναι ε, ο κινητήρας, λέει ο κύριος Κράμερ. Μα από το 2007 υπάρχει ε, απόφαση του Κοινοβουλίου να είναι ελαφρύ πετρέλαιο και όχι βαρύ πετρέλαιο. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο να παραμείνει και να διατηρείται να τηρείται η νομοθεσία. Λοιπόν, ε, συνεχίζω. Μπορεί να είναι εσωτερική ναυσιπλοεία μια πάρα πολύ ε, καθαρή ενέργεια. Ε, για το 2015 έχουμε συμφωνήσει στην Ολλανδία από τότε που ήμουν υπουργό με τον κλάδο να είναι καθαρή η να μην ρηπαίνει δηλαδή η εσωτερική ναυσιπλοεία. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσδοκούμε οπωσδήποτε. Επίσης θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια, σας είπα, σε επίπεδο ερευνητικό. η έξτρα εξυπηρέτηση, το έξτρα handling που χρειάζεται πάντα εσωτερική νευσηπλοεία να γίνει με τρόπο καθαρό, σωστό και χωρίς να αυξάνει πολύ το κόστος. Κάτι που είναι ιδιαίτερα περίεργο. Όλοι ζητούν μεγάλα πλοία και πρόσφατα συζητούσαμε με την Ένωση των Εσωτερικών Λιμένων είχε έρθει και ο διευθυντής τους και κάναμε μια διάσκεψη και ήταν το Colruyt, ε, πώς τους λένε τους άλλους, ε, Arcelor Mittal, οι μεγάλοι πελάτες, ε, μας έλεγαν ότι θέλουν μικρά πλοία. <laughs> Αυτό ήταν πολύ καινούριο για μας, για πρώτη φορά ακούστηκε. Μέχρι τώρα θέλανε να είναι τεράστια τα ποταμόπλια, για να βάζουν πολύ φορτίο. Άρα τώρα φαίνεται ότι αλλάζει η αγορά και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις ανάγκες της. Σε πολλές χώρες οι μικρές διόρυγοι και οι μικρές ε, οδοί ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ποταμόπλια και θα πρέπει να το δούμε αυτό εάν θέλουμε ε, να προχωρήσουμε και με ποιο τρόπο. Να είμαστε πιο αυστηροί κατά των καθυστερήσεων, κύριε Γκρός. Η Συντονιστέ έχουν λόγο, εξουσία δεν έχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα ενδεχομένω. Το πιο δύσκολο εδώ είναι ε, να εφαρμοστεί η ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η περιβαλλοντική νομοθεσία για τους νεοφερμένους στην Ανατολική Ευρώπη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να την εφαρμόσουν και κάναμε μία πρόταση να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων που να δώσει ένα οδικό χάρτη, ένα πρόγραμμα ε, σταδιακής τήρησης και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για να έχουμε και εκεί ε, ένα γνώμονα για το πότε έχουν προχωρήσει και πώς τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλες όντως οι καθυστερήσεις σε αυτό το δομέα. τωρα Τώρα σύστημα 2-2. Σε ή Ζ λέγεται η λεγεται η είναι μια διεθνής ε, γαλλική επιτροπή για να μας συμβουλεύει για, για να συμβουλεύει τους Γάλλους ε, για τα διόδια και περιμένουμε να γίνει και ανάλυση του προβλήματος. Έχει μια έρευνα από το Παρίσι στο Άμστερνταμ για το εξωτερικό κόστος ε, των οδικών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών και μετά θα έρθουν διόδια. Τα μικρά σκάφη όμω, τα οποία ήδη πηγαίνουν στο Παρίσι, φτάνουν μέχρι το Παρίσι, δεν θα πληρώσουν έξτρα διόδια. Α, είναι σημαντικό. Ε, γιατί θα πρέπει στο κάτω-κάτω αυτό είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Θέλουν και οι διοκτήτε των πλοίων ε, και των ποταμών πλοίων να έχουν κάποιο κέρδο. Δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτικό λοιπόν. Για τον Μάρκο Πόλο σα χρωστάω μια απάντηση. Μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια, αν θέλετε και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πολύ σημαντικό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι δύσκολο να στρατολογηθούν, ε, ας πούμε, να βρεθούν στελέχη για τις εσωτερικές πρώτες οδούς ε, που να γνωρίζουν. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν ναυτικοί για τα ποτάμια. Ε, ο κύριος Χαντράουι. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά σας. <laughs> ναι, γελάει ο Σέιντ, ναι. Καθυστερήσεις. Ε, τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να πιέζω τις χώρες καθυστερήσει για τις κυβερνήσεις που αλλάζουν. Ε, αναλαμβάνει μια κυβέρνηση. Εγώ δεν μπορώ να εισβάλλω μες στη χώρα και να πω τι γίνεται εδώ. Ε, χρειάζονται μήνες μέχρι να φτάσουμε στον ε, υπουργό στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω πού. Ε, πείτε να πω ότι κάνετε αυτό, αυτό και εκείνο το, το α και το β στη χώρα σας θα κάνουμε, συμφωνείτε, πώς το βρίσκετε. Δεν θα μου άρεσε αυτό να έρχεται κάποιο στη χώρα μου και να αρχίζει να κάνει διάφορα έργα δεξιά και αριστερά και να μην ξέρω περί πρόκειται. Τι γίνεται με τα διόδια και τους σπόρους. Πηγαίνουν στις δύο χώρες που ε, θα κάνουν τις επενδύσεις, δηλαδή Βέλγιο και Γαλλία. Οι Γάλλοι φαντάζονται ότι θα υπάρχει μια ενιαία επιχείρηση εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα διόδια και θα τα μοιράζει. Οι Βέλγοι λένε, το βελγικό κράτος, ότι ε, θα πρέπει ο καθένας να έχει άλλα διόδια, άλλο τέλος να, πληρω... να καταβάλλεται στο Βέλγιο και άλλο στη Γαλλία. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τομέα. Στρατηγική για το Δούλαβι, η κυρία Μάισνερ, απάντησα λίγο σε αυτό. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, ε, τι γίνεται και εκεί. υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Θα πρέπει ε, τα εμπορεύματα να φύγουν από τις οδικές μεταφορές. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ ε, μίλησε για προσαρμογή των πλοίων στο Δούναβι. Μα το θέμα είναι το μέγεθος των υδατοφραχτών και τα λοιπά. Είναι τεχνικά ζητήματα και αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλη η κίνηση στο Δούναβι. Είναι πολύ λίγα πλοία και τα περισσότερα είναι παλιά, παλαιού τύπου και ρωσικά ε, στην κατασκευή τους. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να γίνει μια διασύνδεση με το Ρήνο. Και θα πρέπει το πλοίο, δηλαδή να ανταποκρίνεται το ποταμό πλοίο και στις προδιαγραφές για την κυκλοφορία στο Ρήνο. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Γκαντσιά, έχετε απολύτως δίκιο. Πολύ καλές ερωτήσεις σας. Η Ιταλία στον Πάδο έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή χωρίς ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση καθόλου. Άρχισαν ε, στη Μάντοβα και είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια που έχουν κάνει και πραγματικά συγχαρητήρια. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ καλές ερωτήσεις και σημαντικές για τη διαλειτουργικότητα. Βεβαίω πάρα πολύ σημαντική και αυτή και θα πρέπει ε, να πετύχουμε. Αυτό είναι το παράδειγμα του Σικουάνα προς τη Βόρεια Θάλασσα το κανάλι, Σεν Νορ. Και ε, μπορούν να διδαχθούν και άλλα έργα αυτά και για το Ρήνο και ε, για, την Ιταλία, για το Δούναβι και για την Ιταλία. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Η επιστολή του Προέδρου της ε, Επιτροπής Παρακολούθησης, ε, τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να ε, επικρίνω τη γερμανική νομοθεσία. Μετά από μια καταγγελία της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέτασα ε, τι έγινε και διαπίστωσα ότι όλα ήταν σύνομα, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία. Δεν είναι δική μου δουλειά να επικρίνω ή να μιλήσω για τη γερμανική νομοθεσία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από πολιτικούς και όχι από την εταιρεία RMD. Και η καταγγελία που ήρθε από την Επίτροπη Παρακολούθησης έχει εξεταστεί. Δεν είναι μόνο από την RMB οι εμπειρογνώμονες και οι σύμβολοι Μπορώ να σας δώσω και την επιστολή να τη διαβάσετε, να μην επεκταθώ σε αυτό. Και στον τύπο δημοσιεύθηκε και δική μου επιστολή. δική μου, που δεν ήταν ακριβώς η δική μου, ενώ δεν ήταν ολόκληρη η επιστολή, γιατί αυτά που γραφική ήταν ακριβώς το αντίθετο των όσων είπα εγώ και των όσων εννοούσα. Ο κύριος Κράμερ, για ε, το Δόναβε μιλήσατε για υδατοφράχτες. Αυτό που θέλει ένας επιχειρηματίας είναι, είναι βέβαιος πόσες μέρες μπορεί ένα πλοίο να περάσει το Δούναβι. Αυτό δεν είναι δεδομένο και δεν έρχονται να επενδύσουν ε, για τη μεταφορά από το Δούναβι γιατί σου λέει δεν είναι πλωτός ε, ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών το χρόνο. Δεν μπορώ να ε, υπολογίζω σε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Βαλιέντ, α, και κάτι που ξέχασα, μια πρόταση. Υπάρχει μια πρωτοβουλία και στην Ισπανία μάλιστα για την εσωτερική ναυσιπλοεία και στην νότια παρακαλώ Ισπανία. Γι' αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη καινοτομία. Οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Επιτρέψτε μου να τις να απαντήσω λακωνικά, προσπαθώντας όμως να καλύψω όλα τα θέματα. Πρώτον, το θέμα της σχέσης με άλλες επιτροπές. Είμαι έτοιμος να πάω σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή, περιφερειακή, περιβαλλοντική, δίχως άλλο είμαι στη διάθεσή τους για να διευκρινίσω τι ακριβώς συμβαίνει με τις θαλάσσιες λεωφόρους και τα άλλα θέματα. Σε ό,τι αφορά το Μάρκο Πόλο και το ΤΕΝΤΙΟ, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε υποβάλει 14 επιλέξιμες προτάσεις. Αυτό έγινε μετά από συζητήσεις. Θα πρέπει να πω ότι αποδίδω μεγάλη σημασία στις επαφές με όσου πρότειναν αυτά τα προγράμματα για αυτέ τι υποψηφιότητε. Θεωρώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή στου παρόντε ισχύοντε κανόνε. Κυρίω κυρίως ό,τι αφορά το Μάρκο Πόλο. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πω ότι εάν υπάρχει εντύπωση ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος, όχι από τις λιμενικές αρχές, Οι λιμενικές αρχές, τουλάχιστον αυτές τις οποίες μίλησα, εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι λιμενικές αρχές, καθώς και όλοι όσοι κινούνται στην ενδοχώρα, εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτού του είδους τα προγράμματα. Η μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι αλήθεια ότι η γραφειοκρατία είναι πολύ πιο εμφανής στους, ε, ε, στα, λιμάνια. Απαιτείται πάρα πολύ σε χρόνο στις διάφορες υπηρεσίες, στην κτηριατρική υπηρεσία και σε άλλες υπηρεσίες για να γίνει η διεκπαιρέωση των διαφόρων θεμάτων. Το καλό όμω είναι ε, ότι το ίδιο σύστημα ισχύει σε αρκετούς λιμένες. Θα μπορούσαμε λοιπόν σταδιακά να προσεγγίσουμε μια κοινή άποψη και μπορούμε να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο γιατί οι διαδικασίες αυτές θα ισχύουν παντού. Εγώ τόνισα το θέμα των logistics δεν είναι αναγκαία τα logistics, η μεταφορά και η αποθήκευση μόνο για τους λιμένες. Είναι απαραίτητη και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επανεξετάσουν τις επιλογές τους. Στις μέρες μας υπάρχει ένα φάσμα υπηρεσιών που συνδέονται με τις μεταφορές Υπάρχει μια φόρμουλα που λέγεται Incoterms και συμπεριλαμβάνει 20 διαφορετικούς τρόπους, 20 διαφορετικές επιλογές που αφορούν τα συστήματα τσίφ και FOB. Είναι πολύ πολύπλοκα αυτά τα συστήματα. Είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς ε, τον ίδιο, το ίδιο των υπηρεσιών που θα μπορούσε να αναλάβουν οι, οι κάτοχοι του φορτίου. Την απόφαση θα πρέπει, του εμπορεύματος, με την απόφαση θα πρέπει να τη λαμβάνουν εκείνοι. Εκείνοι ε, είναι υπεύθυνοι για τα logistics. Βεβαίως το προσωπικό, το λιμενικό προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που εγώ έχω κατά νου είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια γενική βελτίωση της ποιότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η επέκταση του Eco Bonus στο Euro είναι μια καλή ιδέα, υπό τον όρο ότι δεν είναι πολύπλοκο την άποψη των διαδικασιών. Το αρχικό πνεύμα των ε, Ιταλών ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ο οδηγός είναι εκείνο που ε, παίρνει την απόφαση. Θαλάσσια ή χερσαία οδός. Αυτό είναι ένα πολύ ασφαλό, ασφαλές μέτρο σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική πτυχή. Γιατί το ποσό που δίνεται στον οδηγό αντιστοιχεί στο εξωτερικό κόστος του εγχειρήματο. Δεν είναι κάτι ασαφές. Είναι κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί, βεβαίως θα μπορούσε να βελτιωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας συζήτησης θα πρέπει να έχουμε στο νου τη θεωρητική βάση, αλλά και την ταχύτητα. Το πόσο γρήγορα αμείβεται. Γιατί αυτό θα μπορούσε να τον πείσει να περάσει από τις ε, χερσαίες θαλάσσιες μεταφορές. Η ιδέα μου είναι ότι αυτό θα μπορούσε να βρει σύμφωνε και τι μεμονωμένε χώρε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο δύσκολο μέχρι τώρα που διαπίστωσα είναι η συνεργασία μεταξύ των χωρών. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα για το Eurobonus και αυτό αφορά την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Γιατί υπάρχει μια πολύ καλή διασύνδεση μεταξύ της Ιταβέκια και της Βαρκελόνης και αυτή η σύνδεση λειτουργεί πολύ καλά. <clears throat> Είναι λαδωμένα τα γρανάζια και το πράγμα κυλάει. Είναι πολύ καλό το να υπάρχει ένα ε, σύστημα στην Ιταλία όχι στην Ισπανία, όχι στην Γαλλία. Και η Γαλλία θα υποφεληθεί περισσότερο από το σύστημα. Το πιο δύσκολο λοιπόν που προβλέπω ότι θα είναι για το σύστημα είναι το να υπάρξει ένας συντονισμός. Το σύστημα λοιπόν θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό και, ότι, και όχι να είναι ένα σύστημα κατακαιρματισμένο το οποίο θα συμφωνούν οι χώρες μεταξύ τους. Εάν είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ναι, αν θέλετε όμως ε, ε, τελειώστε. Βεβαίως συμφωνώ με την ιδέα το να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ σιδηροδρομικών ε, διαδρόμων και άλλων. Συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα αυτή. Συμφωνώ απόλυτα με τα προγράμματα συνεργασίας που υπάρχουν και που αποσκοπούν σε μια επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Τα κριτήρια τώρα. Τα κριτήρια θα πρέπει να στοχεύουν την μείωση της εντατικοποίησης της χρήσης των χερσαίων οδών. Ήδη μίλησα για την ενιαία φυρίδα <clears throat> και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα νησιά. Οργάνωσα μία συζήτηση, ε, μία συνάντηση των εκπροσώπων από τα ευρωπαϊκά νησιά στη Μαδέρα. Το πιο πολύπλογο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι τα νησιά εισάγουν πολλά, εξάγουν λίγα. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσαμε να βρούμε κάτι άλλο, έναν άλλο τομέα απασχόλησης ε, για τα νησιά. Η Μάλτα, για παράδειγμα, δεν έχει πρόβλημα με τις ε, προμήθειες. Υπάρχει το λιμάνι του Μάσας Λόκ και εκεί παρακάμπτονται όλες οι περιπλοκές, όλες οι δυσκολίες. Δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι απλά τα πράγματα, μπορούν να, γίνονται οι ε, εξαγωγές με μεγάλη ευκολία και αυτό το λόγο έχει κάνει εξαγωγές. Ε. Υπάρχει δηλαδή ένας λιμένας μεταφόρτωσης. Ε. Ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμο το να υπάρχει κάποια πρόβλεψη και για LNG. για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τα 14 αυτά προγράμματα είναι υπό ανάλυση. Πιστεύω ότι τα προγράμματα αυτά στα οποία αναφέρθηκαν είναι πολύ καλά. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με τους σιδηροδρόμους, γιατί εδώ έχει γίνει μια ιδιαίτερη ρύθμιση. Τρεις βασικοί λιμένες, τρεις βασικοί ε, και υδροδρομικές γραμμές στη Ρωσία και ένα νέο ε, εγχείρημα βορρά-νότου Θα πρέπει να πω ότι η Βαλτική είναι πραγματικά ενθουσιώδης σε ό,τι αφορά τις ε, θαλάσσιες λεωφόρους. Και νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Τα μεσογειακά, <clears throat> τα νησιά της Μεσογείου. Επισκέφθηκα την Κύπρο. Η Κύπρος έχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Η Λεμεσός είναι ένα λιμάνι με πολλές δυνατότητες και αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό. Θα πρέπει να τελειώσετε. Λυπάμαι, πρέπει να τελειώσετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρέπει να διακόψουμε. Έχουμε καθυστερήσει 10 λεπτά. Έχω τρεις συντονιστές Κοιτάξτε, αν κάποιος, ε, κάποιο μέλος θέλει μια απάντηση στο ερώτημα που έθεσε, μπορεί να σας ε, ε, την απευθύνει γραπτός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας υποβάλλατε, μας παρουσιάσετε τις εκθέσεις σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της εργασίας σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. call up the next three coordinators.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 Έχουμε πολλά να κάνουμε. Θα πρέπει να περικόψω το χρόνο αγόρευσης. Τόσο απλά τα πράγματα. Θαύματα ξέρω να κάνω. Το μόνο πράγμα που δεν ξέρω να κάνω είναι να ελέγχω το χρόνο. Λοιπόν, θα χρειαστεί να σας ε, περιορίσω το χρόνο, λοιπόν. Right, we'll, we'll get going. We have, όπως γνωρίζετε, έχουμε τον κύριο Ταλίτσκα. Ο κύριος Ταλίτσκα είναι πρώην παίκτη ράγμπι. Βέβαια και εγώ παίκτης ράγμπι είμαι, τώρα δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας είναι ο καλύτερος. Κύριε Στρότσκα, παίζει σε ομάδα των 15 και εγώ στο ράγουμε με τους 13 παίκτες. Λοιπόν, ε, κάντε τις τοποθετήσεις, θα κάνουμε και ερωτήσεις και αν έχουμε χρόνο μπορείτε και να τις απαντήσετε. Παρακαλώ, αρχίστε. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσουμε με τον πρόεδρο ως προς το ράγμπι των 7, το οποίο είναι ε, πολύ ελκυστική ιδέα. Ε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ομολογήσω ότι φέτος νιώθω ότι το έργο μου είναι κάπως πιο εύκολο από προηγούμενες χρονιές, διότι είναι εύκολο όχι μόνο να εξηγήσω και να δείξω την πρόοδο ε, για το θέμα της Βαλτικής, ε, ιδιαίτερα σε ένα διάστημα που ήμασταν ακόμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκπόνησης ε, μελετών, εξέβρεσης συμβιβασμών. Είναι μάλλον δύσκολο να μιλήσει κανείς γι' αυτό και ακόμα πιο δύσκολο να γίνει κατανοητός. Ε, πάντως ε, ήταν ε, πολύ καλό το προηγούμενο έτος για το Rare Baltica και θα ήθελα να πω ότι βλέπω να υπάρχει πρόοδος και όσον αφορά την στάση των διαφόρων κρατών μελών. Ε, αυτό σε εποχή που ε, περνούσαμε δύσκολους ε, οικονομικούς καιρούς που έπληξαν ιδιαίτερα κάποιες βαλτικές χώρες. Πάντως δουλέψαμε καλά, κάποια πράγματα έπρεπε να τα αναβάλουμε. Θα επανέλθω σε αυτό. Έπρεπε να Επιμείνουμε όμως να παραβλέψουμε κάποια ε, ατομικά συμφέροντα και θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ικανότητα κρατών μελών ε, να δείχνουν αλληλεγγύη προς τις γειτονικές τους χώρες. Αυτό δεν το βλέπαμε πάντα στο παρελθόν. Να αναφερθώ τώρα σε κάποια μεμονωμένα σημεία του Rare Baltica να αναφερθώ στα επιμέρους κράτη-μέλη. Η Εστονία για μένα και παρακαλώ μην θεωρήσετε ότι προσπαθώ ε, να κολακεύσω τον ε, ε, επίτροπο που είναι Εστονός. Θα ήθελα όμως να επενέσω την κυβέρνηση της Εστονίας και το Υπουργείο Επικοινωνιών διότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με αναβάθμιση του, της διαδρομής Ταρτού Βάρκα είναι ένα υβριδικό ε, όχημα το οποίο μπορεί να ε, υπάρχει ένα υβριδικό όχημα το οποίο μπορεί να κινηθεί και ε, σε ράγες και στον δρόμο και είδαμε πρόοδο και όσον αφορά την ετοιμότητα του σιδηρομικού σταθμού Βάρκα που είναι πολύ ενδιαφέρον τόπος διότι εδώ βρίσκεται το σύνορο ανάμεσα στις δύο χώρες, ε, την Εστονία και την Λετωνία ε, Ε, ιστορικά όμως ε, κατά καιρούς ήταν ε, πολύ διχασμένοι. Είδαμε λοιπόν βελτίωση στις πλατφόρμες, υπάρχουν, στις αποβάθρες υπήρχαν, υπάρχουν ακόμη κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τους δρόμους αποχώρησης, αλλά φέτος ή του χρόνου η Εστονία θα ολοκληρώσει την αναβάθμιση του δικτύου αυτού. Η επόμενη χώρα που θα αναφέρω είναι η Λετωνία. Εδώ βλέπουμε κάπως ε, το αντίθετο. Είδαμε μια ε, σοβαρή οικονομική κάμψη και οι δυσκολίες που βλέπουμε στη Λετωνία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ε, οικονομική κρίση. Η Λετωνία ζήτησε καθυστέρηση ζήτησε παράταση του χρόνου και μπορούμε να ε, χωρίσουμε την συνδρομική γραμμή της Βαλτικής σε δύο μέρη μέσα στη Λετωνία. Μέχρι την ε, Ρήγα είναι σε καλή κατάσταση, ε, πράγμα που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας των 120 χιλιόμετρων την ώρα για τις μεταφορές. Από την Ρήγα μέχρι τα σύνορα της Λιθουανίας είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Τώρα λοιπόν μετά από τις εκλογές στην Λετωνία ε, λαμβάνουμε κάποια πρώτα θετικά μηνύματα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Στο παρελθόν ε, έχω δει αρκετά θετικά πολιτικά μηνύματα ε, δεν έχουμε δει απαραίτητα όμως ε, αποφάσεις ε, που να στηρίζουν τα μηνύματα αυτά μετά. Ελπίζουμε μέσα στο 2011 να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες, να διατεθούν τα χρήματα ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευαστική εργασία στα τέλη του 2011. Να αναφερθώ και στη Λιθουανία. Η Λιθουανία είναι πάντα πολιτικός πρωτοπόρος ε, όσον αφορά τη συνδρομική γραμμή της Βαλτικής, το Rail Baltica. Ε, υπάρχουν ε, κάποιες δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν. Πιο ενθαρρυντικό και θετικό στοιχείο ήταν η απόφαση το Δεκέμβριο του 2009 να χρησιμοποιηθεί η διπλή ε, γραμμή από, τον, ε, από το πολωνικά σύνορα μέχρι το Κάονας. Γιατί είναι σημαντική η απόφαση αυτή, διότι έχουμε μειώσει σημαντικά το κόστος. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να δημιουργήσουμε ε, νέα γραμμή ε, ε, ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκών προδιαγραφών μέχρι το Κάουνος. Έχουμε λοιπόν την διπλή αυτή γραμμή. Το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο και η ταχύτητα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι μέχρι το 2014 θα έχουμε ε, μέχρι το σε αυτήν την ε, ευρωπαϊκή γραμμή. Και βλέπουμε ότι δημιουργούνται οι τάσεις, η τεχνολογία κινείται γρήγορα, οι αποφάσεις που πρέπει να Σημαντική απόφαση που θα πρέπει να ε, ληφθεί είναι η αυτόματη αλλαγή ε, γραμμών ε, και γιατί το θεωρώ αυτό σημαντικό, διότι αυτό το είδαμε στο παρελθόν και υπάρχουν σημαντικά συμφέροντα εδώ. Είδαμε κάποιες κερδοσκοπικές τάσεις στο παρελθόν αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε αυτόματη ε, αλλαγή του ε, του εύρους των ε, σιδηροτροχιών, διότι η μεταφόρτωση απαιτεί χρόνο, δημιουργεί και ζημιές. Είναι λοιπόν είναι λοιπόν περιττές αυτές οι δυσκολίες. Το άλλο η άλλη σημαντική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες ε, είναι ο σταθμός που θα... Ε, ο σταθμός επιμελητής που θα δημιουργηθεί στο Κάουνας. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα. Κυρίες και κύριοι, να προχωρήσω τώρα στην Πολωνία. Στην ε, Πολωνία ε, βλέπουμε δέσμευση, βλέπουμε ε, ενθαρρυντικά στοιχεία όσον αφορά, αφορά τη γραμμή Βαρσοβίας πλούς και βασικά βρισκόμαστε εκτός των πλαισίων τη ε, χρηματοδότησης, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά το, ε, μέρος, το σημείο περάσματος των συνόρων. Ε, μπορεί δηλαδή να χρειαστεί παράταση για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Εδώ μπορώ μόνο να δεχτώ την προσεκτική, την επιφυλακτική πολωνική στάση που λαμβάνει υπόψη και τις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες ε, θα ε, εκπονηθεί λοιπόν μελέτη για να επιλογεί η σωστή λύση και ε, δεν ξέρουμε αν αυτό θα πραγματοποιηθεί εντός των παρόντων δημοσιονομικών προοπτικών. Πέρσι από τη μία ήμουν επιφυλακτικός, είχα πολλές ελπίδες, από την άλλη ήμουν πεπισμένος ότι ε, θα ε, πετυχαίναμε το όριο των 120 χιλιόμετρων την ώρα. Ε, αν πέρσι λοιπόν ήμουν κάπως επιφυλακτικός, φέτος είμαι πολύ πιο πεπισμένος ότι θα το πετύχουμε. Όσον αφορά την αστυνομική γραμμή Rail Baltica, υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία τα οποία εξετάζουμε. Κάποια στιγμή Ε, είναι σημαντικό να ε, προοδεύσουμε όσον αφορά τις ε, εμπορευματικές, τη διακίνηση απορρευμάτων, διότι αποτελεί το σημαντικότερο όγκο των μεταφορών στη γραμμή αυτή. Σκεφτόμαστε λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να έχουμε υποστήριξη από τα διάφορα κράτη-μέλη για ε, επιβατική γραμμή Ταλίν-Βαρσοβία. ώστε να έχουμε μια τέτοια συνδρομική γραμμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, τώρα είναι κυρίως οδικές μεταφορές. Ε, να μπορούμε δηλαδή να μεταφέρουμε έναν επιβάτη από το Ταλίν στην Βαρσοβία μέσα σε 10-11 ώρες ή αντίστροφα. Ε, αυτό σημαίνει ένα τρένο σε κάθε, κατεύθυνση. Για πολλούς από εμά μπορεί αυτό να θεωρείται αυτονόητο. Αλλά πιστέψτε με ότι στη Βαλτική αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντική εξέλιξη. Ένα τρένο προς κάθε κατεύθυνση και κάποια τρένα ρεζέρβα. Ε, σημαντικό πάντως είναι γίνεται αυτομάτως ε, η αλλαγή του εύρους ε, των, των γραμμών ώστε να μην υπάρχει η καθυστέρηση. Ε, κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν τρένα να λειτουργήσουν με τις προϋποθέσεις αυτές, αλλά αυτό δεν ισχύει ιδιαίτερα στην Ισπανία, το έχουμε δει αυτό και στην Πολωνία το έχουμε δει. βλέπουμε να υπάρχει η δυνατότητα να ε, υπάρχει ε, να γίνεται αλλαγή του εύρους των ε, σιδηροδρομικών γραμμών θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και το απαραίτητο τροχαίο υλικό. ελπίζουμε εντό του χρόνου να έχουμε αποτελέσματα. Αν μου στήσετε συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πολύ δύσκολο να πω κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύουμε μέσα σε δύο-δυόμιση χρόνια ε, να μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα. Το κόστος είναι αρκετά σημαντικό. Έχουμε σημειώσει πρόοδο όμω στη συνομιλή μα με κάποιε εταιρείε. Κύριε Πρόεδρε, ε, πλησιάζω στο τέλο τη παρουσίασή μου. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε. Έχουμε ακόμα κάποιες δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Ε, πιστεύω όμως ότι και με το μνημόνιο που υπογράψαμε πριν κάποιους μήνες έχουμε αρκετά καλή βάση για την δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Επίσης βλέπουμε, και αυτή είναι η τελική μου παρατήρηση, ε, βλέπουμε και κάποια άλλα ενθαρρυντικά ε, σημεία Βλέπουμε το ενδιαφέρον των ε, χωρών της Ασίας, ε, της Κίνας, ε, της Νότιας Κορέας, της Μογγολίας και άλλων, καθώς και κρατών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Βλέπουμε να υπάρχει αυξημένη ζήτηση λοιπόν, ε, βλέπουμε και αύξηση από επιχειρήσεις στην ε, κεντρική Ευρώπη ε, για μεταφορές προς, την, προς τα βόρεια, προς την Πολωνία και κατόπιν ενδιαφέρον για σύνδεση με την Rail Baltica, με τη συνδρομική γραμμή της Βαλτικής. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο μιλητής είναι ο κύριος Σαβαρή, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα προτεραιότητας 22. Ζήλ, καλώς ήρθες και πάλι ε, στο παλιό σου σπίτι. Αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, ε, ζήτησα να μπει ο χάρτης του ε, σχεδίου 22 του Διευρωπαϊκού Δικτύου γιατί είναι 4.300 χιλιόμετρα. Ε, βλέπετε τι είναι αυτό. Είναι οι νέες χώρες διεύρυνσης που με το σιδηρόδρομο συνδέονται. Είναι 160 χιλιόμετρα την ώρα με RTMS ε, ηλεκτρικά και ε, με διπλή ε, ράγα, αν γίνεται, από τη Γερμανία μέχρι την Κωνσταντσα στον Ευξηνοπόντο και περνάει από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και το δεύτερο είναι να απεγκλωβιστεί σιδηροδρομικός πώς η Ελλάδα από τη Βουλγα... και η Βουλγαρία που σήμερα είναι λίγο στο περιθώριο των μεγάλων διευρωπαϊκών δικτύων. Βλέπετε αυτό το χάρτη, το γνωρίζετε ε, και διαπιστώνετε το στάδιο του έργου. Με κόκκινο είναι ε, το στάδιο που δεν έχει αρχίσει καθόλου, κίτρινο αυτό που επίκειται η έναρξη και το πράσινο και το γαλάζιο. Το πράσινο είναι ε, το έργο που έχει ολοκληρωθεί και το γαλάζιο που ολοκληρώνεται. Πολύ πρόσφατα ανέλαβα στη Σαραγώσα, τώρα αρχίζει η αποστολή μου και θέλω να σας δώσω μια ιδέα. 37 ε, ε, ε, ώρες και 23 λεπτά θέλει κανείς από τη Δρέστη να πάει στην Αθήνα και 26 ώρες και 49 λεπτά από τη Δρέστη στη Κωνσταντσα. Χωρίς καθυστέρηση. Το τρένο πηγαίνει με την κανονική του ταχύτητα, έτσι. Ε, γι' αυτό θέλουμε ε, να φτιάξουμε μια σιδηροδρομική γραμμή μικτής χρήσης, εμπορευματικές μεταφορές και επιβατικές μεταφορές. Είναι μεγάλη πρόκληση. Λοιπόν, αν κοιτάξετε το χάρτη εδώ της Ευρώπης θα διαπιστώσετε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στην Τσεχοσλοβακία, λέει ο κύριος Σαβαρή, ε, στην Ουγγαρία, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, ανάμεσα στην Κωνσταντσα και στην Καμπίνα. Ε, βλέπετε τα τμήματα λοιπόν ε, με πράσινο χρώμα που έχουν παραδοθεί και είναι λειτουργικά περίπου στα δικά μας στάνταρ και μετά βλέπετε κάποιες περιοχές πιο περίπλοκες, πιο προβληματικές που είναι η Βουλγαρία ολόκληρη και αυτό το νότιο τμήμα προς την Ελλάδα από τα ουγγρικά σύνορα, Ουγγρο-Ρουμανικά προκειμένου και προσπαθεί να απεγκλωβίσει, είπαμε, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Και υπάρχουν και κάποια μικροπροβλήματα στα σύνορα Τσεχίας-Γερμανίας που από ό,τι φαίνεται εκεί υπάρχουν δυσκολίες και θα επανέλθω να ε, προσαρμοστούν τα εθνικά σχέδια των ε, λόγω κρατών. Λοιπόν, για να δούμε τα θέματα στη γεωπολιτική τους διάσταση περισσότερο. Μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση γενικά δύο ε, ειδών ζητημάτων που απομένουν να λυθούν τα επόμενα χρόνια. Ο πεγκλωβισμος τσεχιας Τσεχίας-Γερμανίας. Είναι δύο οι κλάδοι εδώ. Ο ένας πάει προς τη Δρέσδη, Πράγα-Δρέσδη δηλαδή η σύνδεση και η άλλη είναι Πράγα-Νιρεμβέργη που είναι οι δύο βασικοί κλάδοι του σιδηροδρόμου της σύνδεσης Τσεχίας-Γερμανίας. Οι Τσέχοι σιγά σιγά τελειώνουν το έργο αυτό, το βόρειο τμήμα, Πράγα προσδέστη στα γερμανικά σύνορα ε, είναι στις προδιαγραφές έτοιμο. Και το άλλο τμήμα, στο πούμε ε, νότιο-δυτικό ολοκληρώνεται, δηλαδή Πράγα, Σόντινγκ που είναι τα σύνορα προς τα εκεί. Οι Γερμανοί όμως δεν έχουν ακριβώς τις προτεραιότητες προφανώς ε, σύνδεσης εκεί ε, τα δύο τμήματα των Τζέχων που έχουν τελειώσει. Και η γερμανική κυβέρνηση σαφέστατα έχει σχέδια πάρα πολύ φιλόδοξα και αξιοσημείατα ε, για τρένο υψηλής ταχύτητας. Πράγα, Δρέσδη, Βερολίνο και ε, Πράγα Μόναχο περισσότερο και όχι Νιρεμβέργη μέσω Ρέγγενσπουργκ ή δυνατόν. Αλλά μας λέγουν ότι αυτά τα σχέδια είναι πολύ δαπανηρά σήμερα και ε, δεν μπορούν να εγγραφούν σε ένα ορατό μέλλον. Λοιπόν, έχουμε τα εξή θέμα τώρα. Οι Τσέχοι που βελτιώνουν οι άνθρωποι το δίκτυό τους και απέναντι Γερμανοί που λέγουν μπράβο, πολύ ωραία τα κάνετε, αλλά μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το έργο, γιατί έχω μεγαλύτερε φιλοδοξίε που είναι το τρένο υψηλή ταχύτητα. Αλλά δεν είναι του παρόντο. Έτσι, κάπω δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα, για να μην πω μεγάλη δυσκολία. Πώ αναμένοντα την υψηλή ταχύτητα, ε, περιμένοντα το ICE ε, ε, Πράγα, Ρέγενσπουργκ, Νιρεβέργη, Πράγα, Δρέσδη, ε, Μάλλον, Πράγα, Ρέγγενσπουρ, ε, Μόναχο, χωρί την Ιρεμβερή και κατά τα άλλα συμφωνούν οι Τσέχοι. Λοιπόν, περιμένοντα όλα αυτά, τι θα κάνουμε για να μην ε, ξαναπέσουν όλα στι χερσαίε οδικέ μεταφορέ. Γι' αυτό προσπαθώ, γιατί μου το ζητούν και ενδιαφερόμενοι, κυρίως οι Τσέχοι, ε, να λύσω αυτό το πρόβλημα. Ε, όχι να τους φέρω σε επαφή, έχουν επαφές, αλλά οι Γερμανοί έχουν μάλλον τάση να θέλουν να ε, ε, περάσουν κατευθείαν το βορρά-νότο, βερολινο Βερολίνο-Ρέγγινσπορκ. Και να λένε να έρθουν να συνδεθούν και οι Τσέχοι σε αυτό. Λοιπόν, εκεί είναι ζήτημα. Δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες οι χώρες. Euh, και προσπαθώ να ξαναρχίσω το διάλογο εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει και οι Γερμανοί θέλουν αυτός ο διαδρόμος 22 να μην σταματάει στα τσεχικά σύνορα. Αφού το έχουμε πει ότι θα πρέπει να πάει προς τη Βαβαρία αφενός και από την άλλη μέχρι το ε, λιμάνι του Ροστόκ. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι Γερμανοί γι' αυτό. Να ε, ε, έχει μια διέξοδο. Πράγα Δρέστη, Δρέστη, Λιψία, Λιψία, Βερολίνο, Βερολίνο, Ροστόκ. Εντάξει, δεν λέω θα πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί το σχέδιο, αλλά να ε, καθισκάσουμε τους Γερμανούς γιατί είναι θεμητό αυτό το αίτημα και η προσδοκία. Το δεύτερο τώρα είναι πιο ανισχυτικό. Είναι τέσσερις χώρες του Νότου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή ε, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία. Εκεί μετέβει επί τόπου ε, και στη γέφυρα Βενίν Καλαφάτ και σε όλες τις πρωτεύουσες εκτός από τη Σόφια. Είμαι σε επαφή με την κυβέρνηση. Η μόνη επιτόπου επίσκεψη που μου λείπει είναι η Σόφια. Εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το ποιο είναι το τεράστιο δηλαδή. Οι Ρουμάνοι, το βλέπετε και εσείς στο χάρτη, γεωπολιτικά θέλουν περισσότερο να επικεντρωθούν στον οριζόντιο άξονα, ε, δυτικά-ανατολικά, Ουγγαρία προς την Κωνσταντσα. Απολύτως κατανοητό από οικονομικής πλευράς η προτεραιότητα των Ρουμάνων δεν είναι να βοηθήσουν τον Πειραιά προφανώς και το λιμάνι του θέλουν να ενισχύσουν πρώτα τον άξονα Δύση Ανατολή στη Ρουμανία. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή σε αυτό ε, βάζουν όλες τις προσπάθειες. Στη συνέχεια. Έχουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίε στη Ρουμανία. Οπότε, οι οικονομικές δυσκολίε τους οδηγούν, μεταξύ άλλων, να έχουν και δυσκολίες να ε, συγχρηματοδοτήσουν το εθνικό κονδύλι που τους αναλογεί, οπότε δεν μπορούν απολύτως να απορροφούν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτό αφορά όλες τις χώρες που έχουν τις οικονομικές δυσκολίες, όχι μόνο τη Ρουμανία. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τα, ε, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ακόμα και όταν έχουμε εμείς χρηματοδότηση, δεν μπορούν να βάλουν το εθνικό τους κομμάτι. Και κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει έτσι γενικότερα, όλες αυτές οι χώρες και η Τσεχία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί λένε ότι έχει καταρρεύσει το κλασικό του δίκτυο. Δηλαδή, ε, καταραίει το σύστημα χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου γενικά. Και μα λέγουν ότι έχουμε να κάνουμε τόσα πολλά στον κλασικό σιδηρόδρομο για να ε, κάνουμε μπαλώματα και κάποιε μικρέ γραμμέ, έστω και με 30 χιλιόμετρα την ώρα να λειτουργούν ότι δεν μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητε στα διευρωπαϊκά δίκτυα τώρα ο κόσμο καίγεται. Αυτό μπορεί να μην είναι ευχάριστο να το ακούμε, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε μάλλον... Ε, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνετε ένα τρένο πολυτελεία και να βάλετε όλα τα εθνικά σα λεφτά εκεί. Και τα κράτη λένε «Ε, δεν μπορώ να βάλω τα χρήματα στο τρένο πολυτελεία. Το ξέρω ότι υπερβάλλω, αλλά το λέω επίτηδε έτσι. Ε, και οι χώρε δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να ξυλωθούν εντό εισαγωγικών για το διευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ έχει καταρρεύσει σχεδόν ο εθνικό του σιδηρόδρομο. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ βαριά αυτά τα θέματα και δύσκολα και είμαι πάρα πολύ ανήσυχο, πρέπει να σας πω, για την κόκκινη γραμμή για το νότιο τμήμα, όπου βλέπετε περίπου 6 δις ε, χρειάζονται εκεί, 6 δισεκατομμύρια από τα ουγγρικά σύνορα μέχρι τα ελληνικά ε, και ε, περνάει από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Προς το παρόν ένα τμήμα μόνο, ε, Βιντίν Καλαφά, τη γέφυρα που έχω επισκεφτεί, που 2010 κανονικά θα παραδιδόταν, και στην καλύτερη περίπτωση θα είναι τον Ιούλιο του 2013 με 9 εκατομμύρια ευρώ καπέλο, επιπλέον κόστος. Και εκατέρωθεν θα, ε, μετά τη γέφυρα αυτή το τρένο θα είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή το 2013 θα έχουμε τη γέφυρα αυτή τη Σούπερ και μετά χρειάζονται τρεις ώρες μέχρι την Κραϊόβα που είναι στα 84 χιλιόμετρα από τη γέφυρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο απέχουμε από το στόχο μας. Και θέλω να πω το εξής, γιατί το διαπίστωσα. Ε, δεν είναι ακριβώ θέμα κακής βούλησης προθέσεων των χωρών, γιατί είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η ώρα. Είναι και θέμα ε, διαχείριση, διακυβέρνηση, διασυνοριακής και θέμα χρημάτων. Θα πρέπει να συνεργάζονται οι χώρες και πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλε προσπάθειε για τη διαχείριση, τη διασυνοριακή πλέον αυτών των έργων. Και ξέρετε τι διαπίστωσα, δεν είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα τη διαχείριση, είναι το τεχνικό η καθυστέρηση της γέφυρας Βίντιν Καλαφάτ είναι γιατί έγινε λάθος κατά 50 εκατοστά ε, στη, στο ιδεασμό της γέφυρας γιατί δεν συζητούσανε οι, ε, ε μηχανικοί μεταξύ τους από τη μια Βούλγαρη, από την άλλη Ρουμάνη και δεν συναντήθηκε η γέφυρα ποτέ γιατί έχει 50 εκατοστά απόσταση. Γι' αυτό έχουμε και τρία χρόνια καθυστέρηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα θα πρέπει στα διευρωπαϊκά δίκτυα να ε, υπάρχει μία ε, ε, παροχή συμβουλών, μια βοήθεια τεχνική επιτόπου στον εργοδηγό, στον εργολάβο, δεν ξέρω τι. Όχι υπουργοί, υπουργοί ωραία, υπογράφουν συμφωνίες. η επιμελητή όμως δεν ακολουθεί στη συνέχεια. Ε, για το επόμενο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου των Υπουργών ε, Μεταφορών νομίζω ότι θα ξανασυζητηθεί αυτό το θέμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε ένα κανονισμό που μιλούσε για συμφωνία διακυβερνητική για το 2008 για το κόκκινο τμήμα. Τα χρήματα βρέθηκαν λοιπόν, αλλά δεν προχώρησε το έργο. Το καταλαβαίνει και η Επιτροπή. Προσπάθησαν να το λανσάρω και τουλάχιστον επί τη αρχή συμφώνησαν να υπογραφεί η, διοργανική, η δια, κυβερνητική συγγνώμη, συνεργασία στις 2 Δεκεμβρίου για να μην χαθούν τα χρήματα αυτά. Γιατί θα χαθούν. Και να μην σας πω αν χανόντουσαν τα χρήματα, πού θα πήγαινε αυτό το νότιο τμήμα και αυτό το έργο. Λοιπόν, οι υπουργοί θα υπογράψουν, θα υπογράψουν και οι σιδηροδρομικές ε, ε, εταιρείε και χτυπάω ξύλο, ε, είναι η τελευταία τύχη, γιατί η τελευταία ευκαιρία δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό ε, στη ζώνη αυτή να σκεφτούμε μια ειδική βοήθεια προενταξιακή ε, στα συνδρομικά δίκτυα και στις γραμμές στα Βαλκάνια. Γιατί το λέω αυτό. Διότι δεν είμαι βέβαιος ότι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι θα τελειώσουν αυτό το διάστημα το κόκκινο πριν το 2030. Στην καλύτερη περίπτωση. Το 30 λέω. Στα Βαλκάνια όμως, από το Βελιγράδι, περνούν ε, κάποιες γραμμές που είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα, σε διρόδρομο και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κίνηση και ένα μεγάλο προενταξιακό πρόγραμμα για να απεγκλωβιστεί η Βουλγαρία και η Ελλάδα, ίσως νωρίτερα από ότι να περάσουμε από τη Ρουμανία, που είπαμε η προτεραιότητα της Ρουμανίας είναι οριζόντια. Είναι Ουγγαρία, Κωνσταντσα, οριζόντιος άξονας Δύση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει να πάνε προς τα κάτω. Αυτά, ως μια πρώτη ε, γεύση, μια πρώτη έκθεση για αυτό το έργο που ανέλαβα πρόσφατα στη Σαραγώσα μόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, δεν είμαι, είμαι σίγουρος ότι οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί θα ε, συμφωνήσουν μαζί σας, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ως προς ε, την προτεραιότητα 3, ο κύριος Σέκη, δεν ξέρω αν έχετε εσείς ε, το ίδιο πρόβλημα με τα τούνελ και τις γέφυρες, αλλά θα το ακούσουμε αυτό. Ε, ναι, φυσικά τα ε, διασυνοριακά περάσματα είναι τα πιο ευαίσθητα ε, θα φαντάζεστε όλοι σας πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας. Ε, θα αναφερθώ στην προτεραιότητα 3, όπως είπε ο πρόεδρο σα, ε, αλλά και για το έργο 19. Όπως θα θυμάστε, πέρσι, όταν με όρισαν συντονιστή για την προτεραιότητα 3 μετά τη δουλειά του κυρίου Νταμινιόν που έκανε πολύ καλή δουλειά για την προτεραιότητα 3. Μου ζητήθηκε να είμαι συντονιστής του προγράμματος προτεραιότητας 19, ε, διαλειτουργικότητα στην ε, Ιβηρική Χερσόνησα. Για προφανείς λόγους το θέμα αυτό συνδέεται στενά με το έργο προτεραιότητας 3. Είναι λοιπόν πρώτη φορά που κάποιος ε, σας μιλάει για το ε, δεύτερο ε, έργο και στο έγγραφο που σας έχει μοιραστεί βλέπετε μια γενική περιγραφή του προγράμματος αυτού και όχι μόνο μια επικαιροποίηση. Πρόκειται λοιπόν για δύο πολύ σημαντικά προγράμματα για πολλούς λόγους συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ε, ότι η Ιβυρική Χερσόνησος ήταν αν όχι απομονωμένη, τότε αρκετά απομακρυσμένη από το υπόλοιπο της Ευρώπης όσον αφορά τους ε, συντηροδρόμους. Ε, και για πολλούς τεχνικούς λόγους ε, συνέβαινε αυτό. Ε, ακούσαμε και αυτά που είπε ο κύριος Τελίσκα για την ε, συνδρομική γραμμή της Βαλτικής. Ε, δεδομένων των δυσκολιών είναι πολύ εντυπωσιακή η πρόοδος, η ταχύτητα ανεβαίνει, κοντεύει να φτάσει τα πρότυπα της υπηρετικής Ευρώπης. Ε, βλέπουμε και αλλαγή του εύρου των συνδρομικών ε, γραμμών. Είναι λοιπόν και ένα ενδιαφέρον εργαστήρι ε, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες που υπάρχουν για ιστορικούς λόγους. Όσον αφορά την υψηλή ταχύτητα, το ισπανικό δίκτυο είναι ήδη αρκετά ανεπτυγμένο, όπως ξέρετε, είναι το τρίτο στον κόσμο αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε το 2012 να είναι και το πρώτο εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Πολλές δραστηριότητες λοιπόν πραγματοποιούνται ε, παρότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και δυσκολίες ε, άλλης φύσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Όπως ε, και να έχει και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις ε, καλύτερες ε, συνδέσεις ανάμεσα στην Ιβυρική Χερσόνησο και την Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και όσον αφορά τη ε, μεταφορά με διάφορα μέσα. Επίσης ε, αυτή τη στιγμή ε, βλέπουμε ε, πολύ σημαντικό μέρος των μεταφορών εμπορευμάτων να πραγματοποιούνται στον δρόμο με οδικές μεταφορές, κάτι που προκαλεί συμφόρηση και αποτελεί έναν από τους λόγους που θέλουμε να προοδεύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα με το θέμα αυτό. Υπάρχουν και άλλοι προφανείς λόγοι, η κινητικότητα των ανθρώπων και λοιπά και λοιπά. Και όπως αναφέρουμε και στο έγγραφο που έχετε μπροστά σας, ε, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Να σας δώσω τώρα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να στηρίξω τη δήλωσή μου αυτή. Καταρχήν λοιπόν το PP3, το σχέδιο προτεραιότητας 3, ε, χωρίζεται σε τρία ε, σκέλη από τη Μαδρίτη. Συνδέεται η ε, πρωτεύουσα με την ε, Κασκίλια Λεγόν, την ε, χώρα των Βάσκων και κατόπιν το Παρίσι. Και αυτός είναι ο Ατλαντικός κλάδος ε, για το οποίο θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Κατόπιν ε, έχουμε την ε, Μεσογειακή Οδό, Καταλωνία, Προβυγγία, Παρίσι. Και τέλος έχουμε την ε, διασύνδεση με την Πορτογαλία. Λισαβόνα μέσω Καστήλας, Λαμάνσα, Εστρεμαδούρα και Σέντρο. Και στα τρία αυτά σκέλη βλέπουμε να σημειώνεται πρόοδος στο διάστημα που προσπαθήσαμε να συμμετέχουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, διευκολύνοντας ε, την κατάσταση όποτε ήταν απαραίτητο. Όσον αφορά το ε, μεσογειακό σκέλος θα πρέπει να τονίσουμε ένα επίτευγμα που πραγματοποιήθηκε που πραγματοποιείται τώρα στο τέλος αυτής της χρονιάς ε, αρχή ε, του επόμενου έτους ε, και είναι το πρώτο στάδιο στη διασύνδεση Ιβηρικής Χερσονήσου με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι η διασύνδεση Φιγκεράς Πρεπινιάν και ελπίζουμε σύντομα να λειτουργήσει. Το μεγαλύτερο μέρος της γραμμής Βαρκελόνη-Φιγκεράς και ε, έχει ολοκληρωθεί και η σύνδεση με το λιμάνι της Βαρκελόνης. Ε, ε, πραγματοποιείται δουλειά σε όλο το σκέλος αυτό και και γύρω στο Δεκέμβριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί η γραμμή, όχι οριστικά. μετά όμως από αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τη Λιόν και το Παρίσι. Ε, η γραμμή προς το Μοπέλια επίσης ε, προχωράει. Ε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το 2016 και μελέτες για τη νέα γραμμή Μοπέλια-Περπινιά έχουν ξεκινήσει. Και εδώ μιλάμε για οριστική ολοκλήρωση το 2000, μέχρι το 2020. Αλλά φυσικά μέχρι τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τμήμα της γραμμής που ήδη υπάρχει. Μεσογειακή γραμμή λοιπόν, ε, η Ατλαντική γραμμή ε, ξεκινά ε, στην Γαλλία, προχωράνε οι εργασίες ανάμεσα στο Λατούρ και τον Πορτό και στην Ισπανία ανάμεσα στη Βαγιαλοδολίτη και το Σαν Σεμπάστιαν. Επίσης για το υπόλοιπο τμήμα έχει καθοριστεί η ευθυγράμμιση και έχουμε διάφορα φόρουμ και διασκέψα ε, όπου, έχουν, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Ε, καλό θα ήταν να βρεθεί ε, ένα κοινό μοντέλο για την λειτουργία όλης της γραμμής αυτής. Αυτό αφορά όχι τόσο πολλούς επιβάτες όσο τις μεταφορές εμπορευμάτων και θα ήταν σημαντικό να συνδεθούν μεταξύ τους όλα τα κέντρα διαχείρισης της διακίνησης των εμπορευμάτων ε, στην ισπανική πλευρά. Και η άλλη πρόκληση είναι να καθοριστεί μια πορεία για το διασυνοριακό τμήμα, το, η οποία να ε, ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, αλλά να συμμορφώνεται απόλυτα επίσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή της Ευρώπης. Η Ιβηρική Γραμμή, Μαδρίτη-Λισαβόνα, Περιμένουμε μέχρι το 2013 να έχουμε την ε, πρώτη διασύνδεση ε, υψηλής ε, ταχύτητας μεταξύ των δύο χωρών. Η δουλειά, οι εργασίες συνεχίζονται στην Ισπανία, στην γραμμή 120, 120 χιλιόμετρων, ενώ σύμβαση για σύμπραξη ε, η δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το ε, πορτογαλικό τμήμα υπεγράφει ε, τον Μάιο. Το κομμάτι από τη Λισαβόνα μέχρι την μέχρι τα σύνορα χωρίστε σε δύο μέρη. Για το πρώτο μέρος έχει υπογραφεί η σύμβαση, για το άλλο τμήμα που ε, περιλαμβάνει και το πέρασμα του ποταμού. Ε, υπήρξε σχετική απόφαση η οποία ε, καταργήθηκε και θα επανεφαρμοστεί σύντομα τουλάχιστον ε, με βάση τις ε, διασφαλίσεις που λάβαμε από την κυβέρνηση. Παρότι λοιπόν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και κάποια αναδιοργάνωση εντός της Πορτογαλίας. Ε, ε, ε, περιμένουμε να υπάρξει πρόοδος. Όσοι ήσασταν στην διάσκεψη της Αραγώσας θα θυμάστε ότι προσπαθήσαμε να θεσμοποιήσουμε κάπως τις σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις όχι τόσο για να βελτιώσουμε το πολιτικό κλίμα, αλλά περισσότερο για να έχουμε πιο αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής της δουλειάς μας χωρίς ε, περιττές καθυστερήσεις. Έχει λοιπόν υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των τριών χωρών, ε, Γαλλία, Ισπανία ε, ε, και Πορτογαλία όσον αφορά τα δύο μέρη. Από τη μία θα έχουμε τις σχέσεις ε, Ισπανίας-Γαλλίας και από την άλλη Ισπανίας-Πορτογαλίας. Ε, για το πρώτο κομμάτι θα ήθελα να ανακοινώσω ότι θα γίνει μια τεχνική συνάντηση γύρω στα μέσα Νοεμβρίου για να μπορέσουμε να έχουμε την ομάδα αυτού υψηλού επίπεδου που θα παρακολουθεί την ε, διεξαγωγή των εργασιών. Θα σας κρατήσουμε ενημερούς όσον αφορά ε, το πρόγραμμα 19. Καταλαβαίνω ότι έχω πολύ λίγο χρόνο. Μπορώ κατά βάση να σας πω όμως ότι στην έκθεση θα βρείτε περιγραφή της κατάστασης όσο έχει στους, ε, στις τέσσερις βασικές πορείες Μαδρίτη, Ανταλουσία και στα τέσσερα τμήματα ε, έχει σημειωθεί πρόοδος. Ε, βορειοδυτικά, Μαδρίτη, Λεβάντε, Μεσόγειος και τέλος ε, το, το βορειοδυτικό κομμάτι. Με λίγα λόγια, δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε. Ε, διότι ο πρόεδρος έχει δίπλα του σφυρί του, αλλά για να είμαι σύντομος, νομίζω ότι γενικά μπορούμε να παρατηρήσουμε έντονη δραστηριότητα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις οικονομικές και άλλες δυσκολίες τις οποίες όλοι γνωρίζετε. Πολλά από τα προγράμματα, ιδιαίτερα τα κομμάτια σύνδεσης ε, του δικτύου με τον βασικό άξονα του προγράμματος 3. Στα κομμάτια αυτά λοιπόν βλέπουμε ικανοποιητική πρόοδο. Και βλέπουμε επίσης ε, προσπάθειες να υπερκεραστούν τα προβλήματα στους δρόμους ε, Βλέπουμε όμως ε, και αύξηση της δυνατότητας ε, εκμετάλλευσης του συνόλου της γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δημιουργεί λοιπόν ε, έναν μεσογειακό διάδρομο μεταφοράς πορευμάτων που δεν αποτελεί μέρος του των ε, προγραμματών προτεραιότητας που υπάρχει όμως ε, διότι έχουμε όχι μόνο το πρόγραμμα 3 από την Σαραγώνα ε, προς τα Βόρεια, αλλά έχουμε και το πρόγραμμα 19. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέκη. Η Επιτροπή Μεταφορών του Χρόνου θα επισκεφθεί το κομμάτι Βαρκελόνης-Λιών. Μπορεί να σας συναντήσουμε εκεί λοιπόν. Έχω εννέα βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Τρία λεπτά ο καθένας λοιπόν και θα είμαι πολύ αυστηρός. Θα σας κλείσω το μικρόφωνο αν ξεπεράσετε το χρόνο σας όπως συμβαίνει συνήθως. Δέκα ομιλητές έχουμε. Δύο λεπτά λοιπόν ο καθένας. Δύο λεπτά και ξεκινάμε τον κύριο Κούν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις συντονιστές γιατί οι διάδρομοι και οι διαδρομές από μόνες τους δεν χρησιμοποιούν. Το ζητούμενο είναι το δίκτυο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερα για το σιδηροδρομικό πακέτο για να μπορέσουμε να το επιβάλλουμε και να το εφαρμόσουμε όπως από κοινού το σχεδιάσαμε. Εγώ έχω μια ερώτηση τώρα προς τον κύριο Σαβαρή για το έργο, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο υπαριθμών 22 και μια σύντομη αναφορά στη Γερμανία πώς έχουν καλυφθεί τα ελλείμματα, πώς έχουν κλείσει. Και η γερμανική κυβέρνηση και η ε, γερμανική σιδηροδρομή Deutsche Bahn θεωρούν ότι το Ροστόκ Βερολίνο Κωνσταντσα ε, θα σημάνει ε, κυκλοφορία από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα είναι κονδύλια για τη διευρωπαϊκά δίκτυα εκεί ε, ευρωπαϊκά. Είναι στόχος 1. 160 χιλιόμετρα την ώρα με EMTS θα είναι έτοιμο του χρόνου ε, με διπλή γραμμή για τη ε, διαδρομή, το κλάδο Βερολίνο-Δρέσδη το έχει ζητήσει και ε, η κυβέρνηση της Σαξονίας, η τοπική κυβέρνηση, για να συνδέεται άμεσα η ε, Δρέσδη με το Βερολίνο χωρίς να περνάει από τη λειψία. Και για το Πράγα Νουρεμπέργη ή ε, Πράγα Μόναχο συζητήστε με τον Υπουργό Μεταφορών της Βαβαρίας δεν ξέρω τι θέλουν οι Τσέχοι, αλλά ε, μας, ε, μας ενδιαφέρει στη Γερμανία να συνδέουμε μεγάλα αστικά κέντρα ή μεγάλες περιφέρειες ε, στο διευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ, θα σας υποστηρίξω και εγώ στις διαπραγματεύσεις, αν θέλετε. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και τους τρεις συντονιστές θα ήθελα Κύριε Σίμψον, κύριε Πρόεδρε, να σας ζητήσω το εξής. Και σε σχέση με την εντολή του κυρίου Σέκη. Και... Ε, ε, το βάζει και στην έκθεσή του. Λέει ότι έχει εντολή για να ενημερώνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας. Μιλάω για το σχέδιο 16, έτσι, το διευρωπαϊκό ε, δίκτυο για την κεντρική ε, διάβαση ε, των πυρηναίων. Να μην ενημερώνει μόνο τον Επίτροπο, αλλά και εμά. Γιατί όπως είπε, συνδέεται με το 13 και με το, το 19 συγγνώμη, και το 3 αυτό το διευρωπαϊκό δίκτυο. θέλω να σας πω ότι μας ανησυχούν διάφορα πράγματα η διασυνοριακή σύνδεση του Περπινιάν προχωράει καλά και ξεπερνάει και κάποιες καθυστερήσεις του παρελθόντος με καλό ρυθμό. Και ε, αν είμαι καλώς προφορημένη, νομίζω το Δεκέμβριο θα γίνει η πρώτη διέλευση. Και χαίρεται και ο κύριος ε, Σίμψον, διότι τράβηξε τα πάνδυνα φέτος για να περάσει από το Περπινιάν στην Ισπανία προς τη Βαρκελόνη βλέπω για μια καθυστέρηση ε, τριετίας ε, στην παράκαμψη του Μον Πελιέ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει κάπου αλλού σε συμφόρηση, σε ποτηλιάρισμα. Εσείς εκεί τι προτείνετε. Επίσης είδαμε ενδιαφέρον ε, το, το γεγονός ότι ταυτίζεται ε, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο 19 με τις εμπορευματικές μεταφορές στο σιδηρόδρομο ε, στο διάδρομο της Μεσογείου και χαίρομαι που το είπατε αυτό γιατί δεν ήταν τόσο προβεβλημένο ούτε τόσο ε, σαφές και γνωστό στο παρελθόν. Και τι γίνεται με τη δια, συνοριακή διακυβέρνηση. Καλά τα μνημόνια, καλές οι ομάδες υψηλού επίπεδου. Τι γίνεται όμως εκεί, πώς προχωράει αυτή η υπόθεση στην πράξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, ναι. δύο λεπτά όλοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρώτον, όλα αυτά που έχουν να κάνουν προβλήματα με τη γερμανική κυβέρνηση ε, Είμαι και εγώ πρόθυμη κύριε Σαβαρή να σας βοηθήσω γιατί μας ενδιαφέρει και μας να προχωρούν εκεί τα πράγματα. Το δεύτερο για την προτεραιότητα 3 και 19 κύριε εκεί θα τα αφήσω στους Ισπανούς συναδέλφους μου που ζήτησαν και ίδιο το λόγο της ομάδας μου και αυτά που μας είπε ο κύριος Στήλικα και ο κύριος Σαβαρή ε, είναι προβληματικά και τα γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο. Γι' αυτό ήταν ξεκάθαρο. Κύριε Τσίλικα, είπατε ότι έχει μόνο ε, λεωφοριακή σύνδεση αυτή η γραμμή γιατί πρέπει να αντικατασταθούν οι ράγες οι ίδιες από την αρχή να μπουν καινούριε γραμμές στο σιδηρόδρομο. Και θα ε, είπατε κι εσείς κύριε Σαβαρή, εκτός από τον κύριο Τίλικα. Λοιπόν, ρωτώ, τι απαιτείται για να έχουμε ένα πραγματικό δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη να ολοκληρωθεί, εκτό από τα λεφτά. Εντάξει, λεφτά προ το παρόν δεν έχουμε παραπάνω. Υπάρχει καμιά δυνατότητα να απεγκλωβιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί θέλουμε ένα συνολικό δίκτυο στην Ευρώπη σιδηροδρομικό. Γι' αυτό είναι μεγάλη δυσκολία. Τη Συζητήσαμε και στη Σαραγώσα. Η απλή διασυνοριακή σύνδεση δεν επαρκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ. Καταρχάς πιστεύω ότι γενικά θα πρέπει να απαντηθεί το εξή ερώτημα. Όταν λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα. Η Ισπανία για μένα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δίνει περισσότερα χρήματα για το σιδηρόδρομο από ότι για τον αυτοκινητόδρομο. Όλοι οι υπόλοιποι επενδύουν στον αυτοκινητόδρομο και τελευταίο τροχό τη αμάξη είναι το τρένο. Και στη Γερμανία, σαφέστατα. Και όταν κλέγονται για τα λεφτά, υπάρχει δυνατότητα ε, ε, στα φορτηγά ε, από 3,5 τόνους και πάνω να αυξηθεί το τέλος, το διόδιο σε όλου του αυτοκινητόδρομους. Δεν το κάνουν. Πολύ λίγα κράτη, μόνο η Ελβετία μάλλον γιατί δεν είναι μέλο τη Ένωση. Ε, υπάρχουν λεφτά και βρίσκονται εκεί να τα πάρετε από τον αυτοκινητόδρομο. Οι σύραγγε ε, στον Κοτάρ α πούμε, και αλλού στη ε, Ελβετία χρηματοδοτούνται από τα διόδια που πληρώνουν τα φορτηγά. Γίνεται λοιπόν αυτό. Για το έργο υπαριθμό 17, εγώ πώ το αντιλαμβάνομαι. Το τμήμα ε, στην Πολωνία μέχρι τη Λιθουανία, μέχρι τα σύνορα, ε, επιδιορθώνεται, εξηγένεται και υπάρχουν οικονομικά, οικολογικά προβλήματα. Υπάρχει γραμμή. Εγώ έχω πάρει το τρένο. Για το Κάουνας το καταλαβαίνω ότι θα είναι ένας κόμβος που θα αλλάξει και στην Πολωνία ε, χρειάζεται επίσης αλλαγή. Ε, τώρα από το Δούναβι προς την Κωνσταντσα. Κύριε Σαβαρή, λέτε ότι είναι η προτεραιότητα των Ρουμάνων. Ε, μα αυτό είναι παράλληλο με το Δούναβι. Τώρα μιλάμε για δισεκατομμύρια ε, στο Δούναβι. Ε, θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν. Ε, ή το, ή το σιδηρόδρομο ή το Δούναβι. Χρειάζεται και ένας διάδρομος προς τον Νότο. Και αυτό με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Σερβία ιδιαίτερα το βρίσκω καλό και σωστό και δείχνει και ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον γιατί αν θεωρούν οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να αποφασίσουν και να ε, έχουν τη μόνη σύνδεση προς τον Νότο, να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλη λύση για την Ισπανία. Τι γίνεται με τα Πυρηναία, με τη σύραγγα που θα κόψετε στη μέση τα Πυρηναία, αυτό έχει εγκαταληφθεί, συνεχίζεται. Ξέρουμε ότι στην Ισπανία είναι μεγάλη η προτεραιότητα, είναι πολύ σημαντικό το θέμα, στη Γαλλία όχι. Ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συντονιστές για την πρόοδο που έχει καταγραφεί. Το ερώτημά μου βεβαίως αφορά το σχέδιο για τη Βαλτική. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα, για τα όσα περιγράψετε, καθώ και για το γεγονό ότι είστε πιο αισιόδοξο από ό,τι ήσασταν πριν. Καταρχά, ό,τι αφορά την ε, Λετωνία, τι αναμένετε από την ε, νέα κυβέρνηση, πώς αναμένετε να είναι ε, τα πράγματα. Η κυβέρνηση πάνω κάτω αποτελείται από τα ίδια κόμματα. Το άλλο, το δεύτερο θέμα αφορά την Πολωνία. Έχω ορισμένου προβληματισμούς για το 2013. Τι θα γίνει με την ε, Πολωνία για τον ε, άξονα Έλκα Μπόλαστοκ που θα μπορούσε να επεκταθεί και περισσότερο. Το τρίτο θέμα αφορά τα επιβατικά τρένα. Συμφωνώ ότι και εμείς θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμε τα τρένα μας με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ελπίζουμε του χρόνου να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να υπάρχουν διεθνείς κοινοπραξίες που θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο κατά την άποψή σας θα ήταν το πιο αισιόδοξο σενάριο. κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ ε, ε, σε όλα τα προγράμματα. Ευχαριστώ όλους τους ενδιαφερμένους. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα του Ζήλ Βαρή, του αγαπητού, αλλά μερικά θέματα είναι πιο ενδιαφέροντα για μας. Ε, ο κύριος Σέχη, καλωσορίσατε, είναι σκηταλοδρομία. Τώρα έχετε αναλάβει εσείς τη σκητάλη και κάνετε τη διαδρομή σας πιο γρήγορα και καλύτερα για να είμαστε και δίκαιοι. Ε, εκείνος που δήλωσε, μάλλον και το γεγονός ότι είπατε ότι είστε ε, συγκρατημένα αισιόδοξο και ικανοποιημένο, μα ικανοποιεί και εμά. Αλλά δεν είναι όλα θετικά. Α είμαστε ειλικρινεί. Η κρίση πλήττει του πάντε. Όχι βέβαια τύπου ε, Ρουμανία και Βουλγαρία, όπω είπε ο Σαλβαρή, αλλά μην το ξεχάσουμε. Όλοι έχουμε ένα κοινό σχέδιο. Και τώρα ακούμε για προβλήματα για την Πορτογαλία. Ε, υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς που μπορούν να κάνουν χρηματοδότηση. Ε, γιατί το, το, ο δημόσιος κορβανάς ε, δυσκολεύεται, το ταμείο είναι μείον και δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα. Τα διασυνοριακά προβλήματα τα γνωρίζουμε και ο συνάδελφ, η συνάδελφος Ινέσα Γιάλα αναφέρθηκε σε αυτό. Στο Κώστα Σάρ, ε, η παράκαμψη του Μομπελιέ καθυστερεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να στραφώ κατά της Γαλλίας ούτε να της επιτεθώ, αλλά το είπε και ο προηγούμενος ε, βουλευτής που δεν συμφωνεί πάντα μαζί μου. Ο καθένας κάνει τα καθήκοντά του ε, και τα διασυνοριακά προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε ε, τα δίκτυα να είναι διευρωπαϊκά πραγματικά και να μην ε, σταματούν στα σύνορα. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υπάρχει ο Μεσογειακός Διάδρομος Βέβαια δεν είναι ε, πρόγραμμα προτεραιότητας, αλλά είναι ε, ασυγχώρητο να μην γίνει. Δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ιβηρική Χερσόνησο, για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη Γαλλία. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη πολιτική προσπάθεια και βούληση. Να το κάνετε παρακαλώ. Όχι επειδή θα... Ε, επωφεληθεί η πιο πλούσια περιφέρεια της Ισπανίας γιατί είναι και πολύτιμη συνεισφορά της προς την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και για τη Γαλλία την ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση για τον κύριο Σέκη. Άρχισα να διαβάζω αυτή την διάμεση έκθεση και στη σελίδα 15 αναφέρεται ότι έχουμε καθυστερήσεις Ένας από τους λόγους των καθυστερήσεων είναι οι πολιτικές καθυστερήσεις. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ισπανική και την Γαλλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω θερμά τους τρεις ομιλητές, ιδιαίτερα όμως τον πρώην συνάδελφό μας, τον κύριο Σαβαρή. Ε, είναι πολύ δύσκολο το δικό του κομμάτι, αυτό μπορεί να το πει δικαίως κανείς. Η αξία αυτής της διαδρομής ε, δεν αντιστοιχεί σε αυτήν ε, που τη δίνεται, διότι η σύνδεση αυτή για την οποία μιλήσαμε είναι πολύ σημαντική, διότι ε, μπορεί να συνδεθεί με, ε, με τον Δούναβη τελικά. Έχουμε την τη συνδρομική πορεία από το Λίντς προς τα Βόρεια, ε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σύνδεση με τους τρεις άξονες που αναφέραμε. Ε, είπατε ότι η υψηλή ταχύτητα δεν έχει επιτευθεί ε, στο, στη διαδρομή αυτή και αυτό είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι επειδή μιλάμε κυρίως για γραμμή εμπορευμάτων η υψηλή ταχύτητα δεν θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα. Ήδη δηλαδή με μια επαρκή ταχύτητα θα έχουμε ήδη πετύχει πάρα πολλά. Ακόμα και αν δεν πετύχουμε την τελική υψηλή ταχύτητα, άλλωστε μιλάμε για ορεινές περιοχές, δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει σιδηροδρόμος σε αυτές. Πιο χρήσιμο θα είναι να συγκεντρωθούμε σε θέματα διαλειτουργικότητας και σύνδεσης με τους άλλους διαδρόμους. και την πολιτική στον τομέα αυτόν να την προσανατολίσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Ξέρω ότι ε, οι περιοχές βόρεια από εμά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την διαδρομή αυτή και η Τσεχία έχουν όμως προβλήματα με τις εθνικές κυβερνήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συντονιστές για τα όσα μας ανέφεραν. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σαβαρή ότι συμφωνώ Μένα από τα πράγματα που είπε. Θα πρέπει να υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ε, χώρες μέλη να αντιδράσουν, να κάνουν κάτι εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Το πρόγραμμα 2020 μιλάμε για ηφορία, για ανταγωνιστικότητα και πιστεύω ότι το να επικεντρωθούμε στην εκτέλεση των το προ... προγραμμάτων κατά προτεραιότητα μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ και συμφωνούμε με όσα είπατε γιατί μερικές φορές οι χώρες ε, μέλη δεν το συνειδητοποιούν. Κύριε Σέκη, σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα 3, δηλαδή τις, ε, χώρες, ε, τις βασικές χώρες, Με συγχωρείτε τη χώρα των Βάσκων, πώς θα αξιολογούσαμε αυτά που έγιναν την τελευταία χρονιά. Κατά την άποψή σας, ε, τα πράγματα προχωρούν με τον προβλεπόμενο ρυθμό ή έχουν συσσωρευτεί καθυστερήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τη Γαλλία, είπατε ότι η Ισπανία υπέγραψε τρία μνημόνια. Το σχέδιο όμως αυτό έχει δυσκολίες. Έγινε αναφορά σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Θα επιθυμούσα να γνωρίζω με ακρίβεια πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Η προτεραιότητα 3 προχωράει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Ισπανίας για την ε, χώρα των Βάσκων. Θα ήθελα επίση να γνωρίζω αν λύσαμε το πρόβλημα της σύνδεση με τη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα περί τίνο πρόκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, θα σας δώσω το λόγο αν έχετε τη δυνατότητα σε ένα δεκάλεπτο καθένα να απαντήσετε. Υπάρχουν ορισμένα έγγρα, ε, έργα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ορισμένες χώρες, ε, ε Περπινιών, τη Βερκελόνη ή ε, έργα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Νομίζω ότι εκεί τίθεται το θέμα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από σας, κύριε Τερίτκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τέλος, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα που αφορά τη μεταφορά των επιβατών. Μου είπατε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό. Αυτό θα το αφήσουμε στις μεμονωμένες εταιρείες σιδηροδρόμων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μονοπολιστική συμπεριφορά, προστατευισμός, υπάρχουν συμφέροντα. Ο μόνος τρόπος ε, λοιπόν που μπορώ να φανταστώ είναι το να γίνει μια εταιρεία μεικτών συμφερόντων, να γίνει ένας νέος φορέας ο οποίος θα ασχοληθεί με την λειτουργία αυτών δικτύων. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι θα ξεκινήσουμε πολύ πιο γρήγορα, θα ξεπεράσουμε ορισμένες πολιτικές δυσκολίες, θα ξεπεράσουμε την, ε, μια προσέγγιση που στρέφεται, είναι περισσότερο ε, εθνική, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει μια λογική πίσω από αυτή την ε, ε, ιδέα της κοινοπραξίας. Τώρα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί πρακτικά. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος ε, της ε, χρονιάς θα γίνει πρώτη συνάντηση, χρειαζόμαστε την πολιτική συνένεση και όπως κάναμε και την προηγούμενη χρονιά θα προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα για τη Λιθουανία και για τις χώρες Βαλτικής. Εάν υπάρξει συγκεκριμένο αίτημα βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Πολωνία. Συχνά ακούω παρατηρήσεις για τη μία χώρα ε, σε ό,τι αφορά την άλλη, ότι βραδίνει τα πράγματα. Είναι λίγο παραπλανητικά όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη δέσμευση ε, που αφορά την ε, πλευρά της Πολωνίας αλλά και το τμήμα ε, των σύνορων με την ε, Λιθουανία. Αυτό είναι ένα πρόσκομα πραγματικό. Με ρωτήσατε ε, αν θα μπορούσε αυτή η μελέτη να γίνει νωρίτερα. Η απάντησή μου είναι καταφατική. Ναι, έτσι, έτσι είναι. Βεβαίω το θεμητό ερώτημα είναι εάν θα υπάρξει μία παράκαμψη ή αν θα χρησιμοποιηθεί η πεπατημένη. Εάν κοιτάξετε τα ήδη, τι, τι, τις ήδη υπάρχουσες ε, ράγες διαπιστώνεται ότι είναι γεμάτες ε, ε, στροφές. Από περιβαλλοντική άποψη είναι περισσότερο ε, βιώσιμη. Κύριε Κράμερ, σας ε, απασχολούν τόσο πολύ τα περιβαλλοντικά θέματα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει μία μελέτη σε ό,τι αφορά την ε, Λετωνία. Είναι αλήθεια ότι θα υπάρξουν προβλήματα παρεφερεί με αυτά που αντιμετωπίσαμε ε, πριν από τις εκλογές. Τώρα βεβαίω η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε μια πολύ ισχυρή θέση. Θα χρησιμοποιηθεί όλος ο χρόνος που απομένει για να περατωθούν όλες οι μελέτες και θα ξεκινήσει το έργο το τέλος της επόμενης χρονιάς. Αν δεν γίνει αυτό, είτε είναι η Λετωνία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλη χώρα, θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι θέμα αλληλεγγύης. Εάν δεν συμμορφωθεί ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να ε, κάνει χρήση ορισμένων ε, προνομίων. Τελευταία παρατήρηση που δεν αφορούσε τη Βαλτική, αφορούσε τα διόδια. Ένα ε, ιδιαίτερα σχετικό θέμα που αφορά τη διασύνδεση μεταξύ χερσαίων και σιδηροδρομικών ε, οδών. Δίχως άλλο η χώρα σας θα έχει ένα γενικό σύστημα ε, διοδίων. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα να ακούσω την άποψη του νέου Υπουργού Μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, το θέμα που έθεσε η, ε, ο, κυρία Μάσινε, τι θα πρέπει να γίνει. Η απλή απάντηση είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα όσα έχουν σχεδιαστεί και τα όσα έχουν αποφασιστεί. Δεν ξέρω να υπερβάλλω, αλλά το 1 τρίτο των δαπανών που προβλέφθηκαν το καλοκαίρι αφορούν μελέτες. Αυτό συνεπάγεται ένα μεγάλο όγκο εργασία και ο στόχο ήταν ότι αν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστο, δεν θα έχουμε μια πραγματική διασύνδεση. Διανύουμε δύσκολε εποχέ, εποχή ύφεση και αυτό δεν είναι εφικτό. Καταρχά θα πρέπει να εφαρμοστεί ό,τι είναι εφαρμόσιμο, μετά θα πρέπει να ετοιμαστούμε για τα επόμενα χρόνια και σήμερα θα πρέπει να έχουμε κατά νου δύο θέματα. Μία περαιτέρω αύξηση της ταχύτητας, αλλά να αποφύγουμε το να ξεπεραστούν τα 200 χιλιόμετρα. Από τα 120 εγώ θα περνούσα τα 160. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος. Αυτό και σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα και σε ό,τι αφορά τους επιβάτες. Δεύτερον, και αυτό είναι θέμα πολιτικής η δυνατότητα σύνδεσης ε, του δικτύου της Βαλτικής με την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Το αίτημα αυτό προέρχεται από τα βορειοανατολικά και νομίζω ότι δεν πρέπει να διαπράξουμε τα ίδια λάθη που κάναμε στο παρελθόν όταν είχαμε, αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τα ε, σύντρορα της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης. Το θέμα είναι η διασύνδεση και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε στρατηγικά 20 χρόνια μπροστά. Λοιπόν, άμεση παρουσία, ό,τι είναι να εφαρμοστεί θα πρέπει να εφαρμοστεί και ύστερα θα πρέπει να ετοιμάσουμε όλες τις μελέτες, να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Βεβαίως ε, και το θέμα της χρηματοδότησης είναι θέμα στρατηγικής και το τελευταίο είναι ένα στρατηγικός προβληματισμός που ελπίζω ε, θα ξεκινήσει από την Κομισιόν. Ο κύριος Σαβαρή. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο συνάδελφο. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κούνη και στην κυρία Μάισνερ ότι με του Γερμανού δεν έχουμε προβλήματα, αλλά ε, προβληματίζονται οι Γερμανοί. Και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ θεμητό. Σας το είπα και προηγουμένως και θα πρέπει να καταλάβουμε τι εννοούμε και να είμαστε όλοι σαφείς. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα δημοσιονομικά και τα ε, κράτη τα δυτικά και τα ανατολικά που είναι ακόμα χειρότερο. Ε, ορισμένα κράτη προσπαθούν να επιλέξουν με βάση εθνικά κριτήρια ε, και δίνουν προτεραιότητα και άμεση επιλογή και πολύ βραχυπρόθεσμη στα εθνικά ζητήματα και παραπέμπουν στις καλένδες τα πιο μακροπρόθεσμα. Αυτό το διαπιστώνω παντού ως συμπεριφορά και στα σχέδια προτεραιότητας και στα δίκτυα προτεραιότητας που δεν έχω άμεση εγώ αρμοδιότητα αλλά τα γνωρίζω και στη χώρα μου τα ζω. Λοιπόν, και γι' αυτό προβληματίζει η Γερμανία. Πώς θα συνδεθεί καλύτερα η Βαβαρία ε, ε, με τη Βόρεια Θάλασσα. Δεν είναι θέματα Ανατολής Δύσης μόνο παντού ε, και δεν το βρίσκω πάρα πολύ εύστοχο. Για τη Δρέστη έχετε δίκιο. Τα πράγματα προοδεύουν, αλλά όχι στο διασυνοριακό τμήμα ε, Δρέστη και Τσίν. Αυτό έχει σημασία όμως. Τα 40 χιλιόμετρα από τη Δρέστη μέχρι τη Τσεχία. Η Τσεχία έχει κάνει μεγάλη επένδυση εκεί, έχει φτάσει στα σύνορα και σταμάτησε. Δεν έχει διέξοδο. Και οι Γερμανοί λένε καλά, επειδή κάποια στιγμή θα έχουμε τρένο υψηλή ταχύτητα, δεν επενδύουμε εκεί σήμερα. Μα δύο είναι οι λύσει. Είτε θα επιταχύνει το έργο για την υψηλή ταχύτητα, είτε θα κάνει μια επένδυση για 15-20 χρόνια. Αλλά η αδράνεια δεν είναι επιλογή. Οι Τσέχοι τι να κάνουν, θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Τσεχία που δεν θα βγουν στη Γερμανία. Προηγουμένω ίσω ε, ε, ήταν συγκεχημένοι αυτά που είπα. Α, για τη Βαβαρία, Νιρεμβέργη, Ρέγγενσμπουργκ. Δεν θέλουν ε, να εγκαταλείψουν την Ιρεμβέργη η Γερμανία, αλλά το θέμα είναι πού θα κάνουν τη διασύνδεση υψηλή ταχύτητα με την Πράγα. Στη σημερινή γραμμή ε, που έχουν ε, ανανεώσει οι Τσέχοι, Πράγα, Σέντινγκ, Νιρεμβέργη ή μήπως αυτό που μελετούν τώρα κάνουν Πράγα Ρέγγενσμπουργκ. Και α του Τσέχου να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, οι Τσέχοι συμφωνούν, ε, δεν του νοιάζει. Α επιλέξουν όμω κάτι οι Γερμανοί. Γιατί οι Τσέχοι έχουν ανανεώσει ε, σήμερα ε, το διάστημα Σέγγιν. Και επειδή όμω οι Γερμανοί λένε κάποια στιγμή θα έρθει το τρένο υψηλή ταχύτητα Νιρεμβέργη ή Ρέγγενσμπουργκ, ε, δεν θα κάνουμε διπλή δουλειά τώρα ε, Σέγγιν. Είναι πολύ ακριβό. Ε, μα αυτό πρέπει να λυθεί όμω ω προ τη συνέχεια και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και να γίνει ένας διάλογος τριμερής γιατί οι Τσέχοι κακομύριδες κάνανε με συνέπεια και ευσυνείδητα αυτές τις επενδύσεις και ε, δεν βγαίνει πουθενά αυτή η γραμμή. Και όχι επειδή οι Γερμανοί δεν θέλουν να κάνουν τώρα τίποτα, αλλά επειδή θέλουν να κάνουν κάτι άλλα σε 20 χρόνια. Λοιπόν, για την κυρία Μέισνερ, νομίζω απάντησα για τη γερμανική κυβέρνηση. Παραμένει ανοιχτό ο διάλογο, είναι ειλικρινή ε, και πάρα πολύ ενδιαφέρον και εύστοχο. Μπορεί να φταίει ότι μεγάλο. Αλλά εντάξει, ναι, θα πάω να δω τι περιφερειακέ κυβερνήσει, αλλά δεν θέλω να στριμώξω την κεντρική κυβέρνηση. Γιατί οι διαπραγματευτές, οι συντονιστές συγγνώμη, δεν διαπραγματεύονται απευθεία με τι περιφερειακές κυβερνήσει. Αλλιώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ε, νομιμότητας. Δεν θα πρέπει να στριμώχνουμε τις κεντρικές κυβερνήσει. Ξέρω ότι υπάρχουν τοπικά προβλήματα και εγώ είμαι πολιτικός τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ε, θέλω πάρα πολύ ε, προσεκτικός εδώ γιατί μπορεί καμιά φορά να βραχικυκλώνουν τις κεντρικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές αρχές και να συνδιαλέγονται με την Ευρώπη απευθεία. Λοιπόν, ε, προβλήματα χρηματοδότησης και του κλασικού δικτύου. Ε, η ε, απελευθέρωση κανονικά ρίχνει το κόστος, αλλά δεν είναι το μόνο, εργαλείο, το μόνο μέσο. Συγγνώμη. Δεν είναι... Κύριε Κράμε, το θέμα να βγάλουμε λεφτά από άλλα μέσα για να πάνε στο σιδηρόδρομο. Οι επενδύσεις στο σιδηρόδρομο είναι βαριές ε, και είναι πολλές γενιές. Ε, είναι κρατικές επενδύσεις, μπορεί να είναι πολλά χρήματα, αλλά τελικά ε, διαρκούν 100-200 χρόνια. Κύριε Κράμερ, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιλέξουμε το Δούναβι ή το σιδηρόδρομο. Πρώτον, ο Δούναβις είναι μόνο εμπορευματικές μεταφορές, δεν θα μεταφέρει επιβάτες να δούμε αν είναι περισσότερο χρήσιμο ο δούναβη επιπλέον του τρένου για τι εμπορευματικέ. Αλλά οι Ρουμάνοι, σας λέω, θέλουν να κάνουν τη γραμμή Ουγγαρία-Κωνσταντσα. Χρόνο θέλουν, λεφτά δεν έχουν πολλά. Είναι δύσκολο, αλλά αν κάνουν κάτι στο έργο, σε αυτό το ε, πρόγραμμα προτεραιότητας 22, Ε, και ε, κυρία Λίχτμπεργκερ, ε, ε, Λίντς Πράγα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. 300 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να βάλει η χώρα σας το χρόνο του χρόνου για το Σούμεραου. Οι Τσέχοι προχωρούν, όλοι συμφωνούν και λέγουν ότι η γεωγραφία, η τοπογραφία, τα τοπία είναι πάρα πολύ όμορφα και θα ήταν πολύ μεγάλο το κόστος αν θέλαμε να κάνουμε ε, γραμμή υψηλή ταχύτητας. Λοιπόν, θα τη βελτιώσουμε για να μεταφέρει εμπορεύματα με τρόπο πολύ πιο άνετο, αλλά δεν υπάρχει η ίδια φιλοδοξία ε, όπως ε, στη Γαλλία, στι ακτέ του Ατλαντικού ή στην κοιλάδα του Ροδανού. Αυτό τώρα που μας απασχολεί είναι πώς θα βγουν στη Μεσόγειο αυτέ οι χώρε. Να περνάνε όλοι από τον Μπρένερ, από τη Σύραγγα ε, ή απαλού. Πολλές είναι οι ε, απαντήσεις εδώ για τους άξονες βορρά-νότου το χώρο της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό μπορώ να σας πω και ελπίζω να έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που θέσατε και για τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να δώσω ορισμένε απαντήσεις. Καταρχάς, το θέμα των πολιτικών καθυστερήσεων. Ελπίζω να μην χρησιμοποίησα λανθασμένα αυτό τον όρο. Αυτό που είπα αναφερόταν περισσότερο σε καθυστερήσεις και πολιτικές δυσκολίες. Αυτό δεν αποτελεί κριτική εντός, ε, ε, ε, προς αυτούς που δουλεύουν με το θέμα, αλλά δείχνει τις δυσκολίες στις διασυνοριακές συνδέσεις. Όταν μιλάμε για διάφορα επίπεδα υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις, ο χρόνος περνάει γρήγορα και αυτός είναι ο λόγος που Ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι που πετύχαμε υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης στη Σαραγώσα. Χαιρόμαστε που θα γίνει και συνάντηση μέσα Νοεμβρίου για να ε, λειτουργήσουν οι ομάδες υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά απαιτούν μόνιμη παρουσία και όπως είπε και η κυρία Αγιάλα Σέντερ, ε, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική βελτίωση. Οι καθυστερήσεις, η έλλειψη χρόνου μπορεί να αποτελούν δικαιολογίε σε πολλές περιπτώσεις που δεν είναι κανείς έτοιμος ή που δεν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις αλλά ελπίζω να μην είμαι υπερβολικά αφελής ε, αν πω ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να ε, συγκεντρώνει κανείς ε, όλα τα μέρη και έτσι συχνά περνάει ο χρόνος υπερβολικά γρήγορα. Αυτή είναι η γενική ιδέα και ε, αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της διακυβέρνησης. Στην πράξη θα δούμε πώς αυτή η πρώτη προσπάθεια που αφορά τη Γαλλία και την Ισπανία θα λειτουργήσει. Λιγότερο με ανησυχεί η Ισπανία, υπόθεση Ισπανία-Πορτογαλία. Θα προσπαθήσουμε όμως και εκεί να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Όπως και να έχει, οι επαφές με ανθρώπους στην κυβέρνηση και σε άλλα επίπεδα είναι μόνιμες και ε, πραγματοποιούνται με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Ωραία. Προτεραιότητα 16. Βεβαίω δεν είμαι εγώ εκείνο που θα αποφασίσει ποιο θα πρέπει να ασχοληθεί. Καταρχά ε, θα σας δώσω μία αγραφειοκρατική άποψη. Αν κινούμεθα στο γενικό πλαίσιο των προτεραιοτήτων, ισχύει αυτό που είπα και στην αρχή. Ότι υπήρχε, υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι για να γίνει για να υπάρξει αυτή η προτεραιότητα. Αυτή είναι η γραφειοκρατική άποψη. Προσωπικά πιστεύω ότι έχει νόημα να αρχίσουμε να δουλεύουμε με βάση ένα παρεμφερές πρόγραμμα που είναι πολύπλοκο, χρειάζεται χρόνος, είναι μακροπρόθεσμο. Αλλά επειδή εγώ ίδιος προέρχομαι από την περιοχή των ε, Άλπαιων. Ξέρω πόσος χρόνος χρειάστηκε για τις σύραγγες, πόσος ε, ε, κόπος χρειάστηκε για να γίνουν. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σκόπιμο να γίνουν προκατακτικές μελέτες ή δυνατόν για να υπάρξει και πάλι η παλιά σύνδεση μεταξύ της Γαλλίας και της ε, Ισπανίας. Ξέρω ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, αλλά ενδεχομένως αυτό θα παρουσιάσει και κάποιο τουριστικό ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση είναι ένας τρόπος για να προχωρήσουμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια για να ξεκινήσουν οι προκατακτικές μελέτες και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε κοιτάζοντας την ενδιάμεση έκθεση που έχετε μπροστά σας υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν αυτά τα χρήματα. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα πρέπει να συνεχιστούν, να προχωρήσουν αυτό το θέμα θα το αναφέρουμε στις δύο κυβερνήσεις όταν συναντηθούμε, απλά και μόνο για να τους θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος και συνήθως θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Τώρα, μεσογειακός διάδρομος. Από το 14 περάμε στο 19. Ο μεσογειακός διάδρομος, όπως είπα, δεν αποτελεί μέρος ενός μιας προτεραιότητας, αλλά τα στοιχεία του είναι τέτοια που είναι σαν να ήταν μέρος ενός τέτοιου προγράμματος γιατί είναι ένας διάδρομος ε, για εμπορεύματα, ε, γιατί έχουν αναπτυχθεί διάφορες παράκτηρες γραμμές από την Ισπανία. Όλοι είμαστε της άποψης ότι είναι μια καλή ιδέα να συνδεθεί καλύτερα όχι μόνο η Βαρκελόνη αλλά και άλλα μεσογειακά λιμάνια. Τίποτα δεν χρειάζεται να προσθέσω. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα συμβεί όταν επαναπροσδιορίζεται μία πολιτική και κυρίως όταν επαναπροσδιορίζονται τα λεγόμενα κεντρικά δίκτυα. Εάν επιτευχθεί μια συμφωνία τότε ο μεσογειακός διάδρομος θα πρέπει να αποτελέσει μέρος του core network, αυτού του δικτύου που συμπεριλαμβάνει πολλά στοιχεία και συμπεριλαμβάνει και αυτό που ονομάζεται μεσογειακό διάδρομο που είναι βασικά για εμπορεύματα και που εν μέρη βρίσκεται σε λειτουργία. Νίμα Μοπελιέ αποφασίστηκε να υπάρξει μία αναβολή για διάφορους λόγους, οικονομικούς, τεχνικούς και λοιπούς. Θα πρέπει λοιπόν να το καταγράψουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση η παλιά γραμμή δεν θα είναι έτοιμη πριν από το 2020. Τα καλά νέα στην περίπτωση αυτή ότι η πρώτη φάση του προγράμματος θα συμπεριλάβει την αύξηση της, ε, ε, του, δυναμικού της υπάρχουσας γραμμής. η σύραγγα του Περπινιάν Φιγέρας δεν θα είναι, όπως λέμε στα Ιταλικά, ε, ένας καθεδρικός ναός μέσα στην έρημο. Σε κάθε περίπτωση Πιστεύουμε ότι όταν το τζεβέ θα φτάσει στο σταθμό το Φιγέρας φτάνει από πολύ μακριά. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουσα γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα ίδια υπάρχοντα. Τέλος. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο του Ατλαντικού, το θέμα που έθεσε η κυρία Μιλμπάο, μολονότι έχουν καταγραφεί καθυστερήσει σε ορισμένα μέρη, η εκτέλεση του κομματιού στην Ισπανία προχωράει Το πρόβλημα είναι το τι θα γίνει στην διασυνοριακή περιοχή. Η Γαλλία είναι σχεδόν έτοιμη γιατί όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από την άφηξη στα σύνορα βρίσκονται σε φάση εφαρμογής. Συνεπώς, το εξετάζουμε το πρόβλημα από την περιοχή της περιφέρειας Ακιτένα όταν τα περιθώρια στερεύουν και όταν η λύση βρίσκεται μπροστά μας. Στη χώρα των Βάσκων τα πράγματα έχουν διευκολυνθεί. Σε κάθε περίπτωση η χώρα των ε, ο σύνδεση των Βράσκων Γαλλίας ε, έχει περιβαλλοντικά προβλήματα. Εδώ θα πρέπει να εξεταστούν διάφορα θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι η διακυβερνητική συνδιάσκεψη έχει τώρα πλέον στη διάθεσή της τα απαιτούμενα για να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα ερεθίσματα από αυτή την άποψη, έτσι ώστε να μην υπάρξει σπατάλη χρόνου. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στα ερωτήματα που ετέθησαν. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Well, can I... σας ευχαριστώ που πήρατε το λόγο. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε στις διάφορες ερωτήσεις. Όπως είπα και στον κύριο Βαλέντε και την ε, κυρία Πέστα, θέλαμε πραγματικά να συνεργαστούμε στενά μαζί σας. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, κυρίως με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όπως σας είπα όμως, εμείς βρισκόμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και αν ε, επιθυμείτε για να γνωμοδοτήσουμε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέσατε και ας δείξουμε την ε, εκτίμησή μας στο πρόσωπο των ομιλητών, αγαπητά μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιστρέφουμε στις 3 και θα ακούσουμε τον Επίτροπο στις τέσσερις, θα τελειώσουμε τους συντονιστές. Θα έχουμε τέσσερις συντονιστές σε μια μισή ώρα. Με τη βοήθειά σας είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Τέσσερις. Όχι, τρεις, τρεις για τον Επίτροπο και τέσσερις για, την, για τους υπόλοιπους και του συντονιστέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη.